Okay, colleagues, I'm going to start the meeting because it is, has actually gone three o'clock. And um, first of all, there is the draft agenda. I think... Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, μάλλον θα έχετε προσέξει πως έχει αλλάξει η ημερήσια διάταξη από το αρχικό σχέδιο, οπότε θα το διατρέξω λίγο. Έχουμε την έκθεση της κυρίας Τσικάου, η οποία δεν θα συζητηθεί σήμερα, οπότε περνάμε στα σκάφη αναψυχής μετά σιδηροδρομικός χώρος, προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και στρατηγική του Ατλαντικού και στις 6 ώρα συντονιστές. Αύριο, μετά τις ανακοινώσεις, έχουμε την ψηφοφορία για τα σκάφη αναψυχής. Μετά η ανακοίνωση των διαπραγματεύσεων για την ΕΜΣΑ και η ακρόση για το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Δεύτερη συνεδρίαση με την Ήτρα στην άλλη πλευρά, στην αίθουσα PHS 3C50. Και το απόγευμα, ξανά σε αυτή την αίθουσα, ανταλλαγή απόψεων με τον ε, κύριο Γιάρζεμπόφσκι και κοινή συνάντηση με την ΙΜΚΟ και μετά παρουσίαση της ε, διαρθρωτικής πολιτικής. Πρέπει να τα ξέρουμε αυτά. Να ξέρουμε πως σήμερα, δηλαδή, να το έχετε κατά νου. Συνεδριάζουμε εδώ, αύριο μέχρι τις 10 και 4 εδώ, μετά πάμε στην 3 σε 50 και μετά το απόγευμα αύριο ξανά εδώ πέρα πέρα δόθε στο κτίριο. Δηλαδή να γυμναστούμε κιόλας λίγο αύριο αυτά. Ε, ζητώ συγγνώμη, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ημερήσια διάταξη. Συμφωνείτε όλοι με την ημερήσια διάταξη όπως ε, είναι τώρα. Ε, και αν πείτε όχι θα την ψηφίσουμε, αυτό θα γίνει. Και αν εξακολουθείτε να λέτε όχι, δεν ξέρω. Μετά δεν ξέρω. ρωτήσω εδώ πέρα αυτούς που ξέρουν τον κανονισμό. Εντάξει. Όλοι ικανοποιημένοι έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης. Ε, συμφωνούν όλοι. Της 26 και 27 Μαρτίου. Ωραία. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην έκθεση Τσίλε. Αλλά ο κύριος Τσίλε απουσιάζει. Well, I think they've just finished the so... Μάλλον θα τελείωσε μόλις τώρα ο τριμερής διάλογος. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς τον εισηγητή μάλλον. Θα περιμένουμε λίγο.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 Λοιπόν, περνάμε λοιπόν στην έκθεση σκάφη αναψυχή και ατομικά σκάφη, εξέταση των τροπολογιών. Κύριε Τσίλε, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους κατέθεσαν τροπολογίες. Συνολικά έχουμε 16 τον αριθμό. Πρώτα απ' όλα, ποιες μπορώ να στηρίξω ή υπαριθμών 16 που ξεκαθαρίζει το κείμενο και την οδηγία. Πρέπει να διευκρινίσουμε τον, το τι σημαίνει εδώ πέρα αμφίβιο σκάφος, γιατί οι σκανδιναβικές χώρες υπάρχουν σκάφη που λειτουργούν και σε, πάνω στο νερό και πάνω στον πάκο και πρέπει να συμπεριληφθούν. Επόμενο, κατοθετικό, είναι η τροπολογία 11 απέτηση στους εισαγωγείς να δίνουν τα απαραίτητα έγγραφα που να περιέχουν το όνομα και τη διεύθυνσή τους. Και η 14 για τον καθορισμό των υπηρεσιών στα κράτη-μέλη που θα εφαρμόσουν αυτή την οδηγία και θα επιβάλλουν ποινές για παραβιάσεις της νομοθεσίας. Επίσης υπάρχουν κάποιες τροπολογίες ε, τις οποίες ε, δεν θα ήθελα να υποστηρίξω προσθήκες στο κείμενο και που μπορούν να μας οδηγήσουν σε κάποια παραπλανητικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα οι 9, 12 και 19. Οι 18 για πιο περιοριστικά μέτρα για τη χρήση προσωπικών ε, ε, ατομικών σκαφών. με επαναλαμβάνει το άρθρο 5 που, το οποίο λέει συνέχεια τα σκάφη αναψυχή και τα ατομικά σκάφη. Δεν προσθέτει τίποτα. Τώρα οι 25 και οι 23. Θέλω συνάδελφοι εδώ να προσέξουν λίγο για τις νέες απαιτήσεις ασφαλείας ε, για τα σκάφη αναψυχής. Ε, είναι βασικό στόχος τη οδηγία Βεβαίως, αλλά πρέπει να φροντίσουμε πως οι προσθήκες οι οποίες προτείνονται δεν καλύπτονται ήδη από τις υφιστάμενε απαιτήσει και ποιε είναι οι φυκτές τεχνικές λύσεις για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσει. Συγκεκριμένα, για την 22, για την προστασία των κολυμβητών, για ορατότητα από την θέση του τιμονιέρη, Υπάρχει ήδη προδιαγραφή ISO και μην ξεχνάμε πως ε, τα περισσότερα από αυτά τα ατυχήματα σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα και όχι με το σχέδιο του σκάφου. Και σημαντική εδώ πέρα είναι οι εθνικοί κανόνες ε, ε, επιχείρηση και χρήσεων σκαφών έτσι ώστε οι περιοχέ κολύμβηση να είναι προστατευμένε ζώνες και να υπάρχουν σαφείς περιορισμοί για τη χρήση των σκαφών αυτών. Επίσης για το 23. Ευχαριστώ να ακούσουμε τα σχόλια τη Κομισιόν γιατί 23 αφορά την περαιτέρω διευκόλυνση επανεπιβίβαση και καλύτερη προσέγγιση από τα άτομα που βρίσκονται μέσα στο νερό. Θέλω εδώ πέρα η Κομισιό να μας εξηγήσει τις υφιστάμενες απαιτήσει, ε, τι σημαίνει, ποιε είναι για την επανεπιβίβαση και να μας δώσει την αποψή της για το εάν ε, είναι τεχνικά εφικτές και θα έχουν τις επιθυμητές ε, βελτιώσεις. Και με τα 24 έως 28 τροπολογίες όλες των πρασίνων για πιο περιοριστικά όρια του θορύβου όπως συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά και έχει γίνει και έρευνα από την Κομισιόν. Ε, απαιτήσει για, τις, για τους κινητήρες για το σχέδιο του σκάφους και τα κοστίζουν πάρα πολύ κοινωνικά και οικονομικά Γι' αυτό θέλουμε οι απαιτήσει αυτές να μείνουν σύμφωνα με την πρόταση της ε, Κομισιόν. Και τέλος η 13 και οι 20 για τις ε, ε, εξουσιοδοτήσεις προς την Κομισιόν. Όχι, πρέπει να παραμείνουν αυτά στην κανονική νομοθετική διαδικασία, την συναπόφαση. Οπότε και οι δύο τροπολογίες δεν ε, στηρίζονται, δεν μπορώ να τις στηρίξω εγώ. Παρά το ότι Ε, δεν ξέρω οι πράσινοι τι επιθυμούν, γιατί εδώ πέρα θα υπάρξει μείωση αυτών των απαιτήσεων. Αλλά εγώ προτείνω την τακτική νομοθετική διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ασάντα για το ΕΛΚ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Μιλάω εκ μέρου του κύριου Μάρτσιν Κέμπιτ, που είναι σκιώδη εισηγητή μα. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε μαζί και για την δυνατότητα να καταλήξουμε σε κοινέ λύσει. Όπω επίση τον ευχαριστώ επειδή έχει καταλάβει και πόσο περίπλοκο είναι το θέμα. Θα σχολιάσω πρώτα τι προτάσει που έχει υποβάλει ο ίδιο εισηγητή. Όπω πολύ σωστά υπογραμμίζει, τίθεται θέμα εκπομπών, επιπέδων εκπομπών ε, και επιπέδων θορύβου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να οργανώσουμε τις προδιαγραφές ασφάλειας του τομέα αυτού. Συμφωνώ λοιπόν με τον εισηγητή για το ότι τα όρια εκπομπών είναι εφικτά. Ιδιαίτερα τα τρία στοιχεία. Και για το διοξίδιο του άνθρακα και όσον αφορά τον θόρυβο. Έχουν υποβληθεί τώρα κάποιες τροπολογίες για τα όρια, αλλά νομίζω ότι οι προτάσεις που υπάρχουν είναι παρκής. Επιπλέον περιορισμοί και απαιτήσει, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας, πιστεύω ότι δεν αιτιολογούνται. Δεν δικαιολογούνται. Πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν ε, και οι μικροί ε, κατασκευαστές και ότι τρία χρόνια περίοδος χάριτος για μικρές επιχειρήσεις είναι κάτι που δικαιολογείται απόλυτα. Ο σκιώδης συζητητής μας επίσης υπογραμμίζει ότι στην τροπολογία 10 θα έπρεπε να κοιτάξουμε το ειδικό καθεστώς των μικρών και μεσαίων ε, επιχειρήσεων. Μια που δραστηριοποιούνται πολύ στον τομέα αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ώστε να επανακτήσουν το κομμάτι της αγοράς που είχαν πριν την κρίση. Εμείς θα προτείνουμε προφορικές τροποποίησεις. Στην τροπολογία 9, για παράδειγμα, θέλουμε να διαγραφεί ο όρος περιβαλλοντικό. Επίσης, πρέπει να αλλάξει και η τροπολογία 10. Ο κύριος Μαρσινκέβιτς προτείνει να χρησιμοποιήσουμε τον όρο επιπλέον, in addition to. Πάντως ευχαριστεί πολύ για το θέμα των βέλτιστων πρακτικών είναι κάτι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να πετύχουμε κοινέ προδιαγραφές. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες και οι ιδέες ε, για τα υβριδικά. Για τις υβριδικές εγκαταστάσεις. Ευχαριστή πολύ επίσης για τις προτάσεις του εισηγητή, τις οποίες βρίσκει γενικά θετικές, αλλά πιστεύει ότι μερικές φορές είναι υπερβολικά περιοριστικές, κάτι το οποίο δεν το βρίσκει σύμφωνο. Καλώς. Ε, ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σπύρος Νανέλης που παρακολουθεί το θέμα αυτό μου είπε πως δεν μπορεί να είναι εδώ πέρα σήμερα, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη γραμμή του εισηγητή διαπιστώνουμε πως ο εισηγητής ε, στηρίζει τις δύο τροπολογίες που κατέθεσε η ομάδα μας. Στηρίζουμε επίσης τον συνάδελφο Ζήλε στην απόρριψη ορισμένων τροπολογιών ε, συναδέλφων που θέλουν να αλλάξουν το τεχνικό παράρτημα της πρότασης της ε, Κομισιόν και να αλλάξουν έτσι, να αυστηροποιήσουν τα όρια του θορύβου. Θεωρούμε πως τα ανώτατα όρια που ισχύουν είναι ικανοποιητικά και έχουν τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να τα κάνουν ακόμη αυστηρότερα. Για να συντομεύω λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Είμαστε ικανοποιημένοι με τη δουλειά του κυρίου Ζήλε και στηρίζουμε την ε, έκθεσή του. Thank you very much. Next is Mrs. the Liberal. Η κυρία Σάλης εκ μέρους των Φιλελεύθερων έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τα σκάφη αναψυχής και η σχετική οδηγία είναι νομίζω κάτι αρκετά ευρύ. Ο εισηγητής έχει πραγματικά αναλύσει και το κείμενο και τις τροπολογίες. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Θέλω όμως να ευχαριστήσω τον εισηγητή πρώτα απ' όλα για τις τροπολογίες του. Στηρίζω τη θέση του εισηγητή και της Επιτροπής για το ότι οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Κάτι τέτοιο βοηθάει τους ε, παραγωγούς. Έρχομαι τώρα στις τροπολογίες. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, όλες οι ομάδες στηρίζουν τις τροπολογίες του εισηγητή για τις υβριδικές τεχνολογίες, τις νέες τεχνολογίες που πρέπει να προωθηθούν όπως επίσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών μελών, είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό. Όπως όμως και οι προλελήσαντε, δεν στηρίζουμε τις τροπολογίε που έχουν να κάνουν με την ηχορύπανση. Γιατί αυτό θα σήμαινε μεγάλες αλλαγές για τους κατασκευαστές. Θέλουμε να περιοριστούμε στα μικρά σκάφη και στην ταχύτητα. Δεν θα πρέπει να υπάρξουν νέοι περιορισμοί. Ούτε στηρίζουμε και τις τροπολογίες για τον σχεδιασμό. Υπάρχουν ήδη κανόνες από τα κράτη-μέλη από αυτού. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την τόσο καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Ζανόνκα από εκ μέρους των Πρασίνων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την δουλειά του, για τη θέση του και για την γραμμή που γενικά στηρίζουμε. Ελπίζουμε οι τροπολογίες αυτές που βάζουν σε κατηγορίες τα σκάφη θα διευκολύνουν την κατάσταση. Όσον αφορά τώρα το κόστος, δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει επιπλέον κόστος. Αυτή είναι και η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι είναι εφικτό να γίνει μείωση του ήχου που προκαλούν το, τα σκάφη, τα 40 κιλοβατόρων κατά 5 τεσιμπέλ. Είναι εφικτό αυτό. Έχουμε βέβαια τη δικιά μας επιχειρηματολογία όταν ε, καταθέτουμε την τροπολογία 22 για τον ε, σχεδιασμό. Μπορούμε, πιστεύω, να βασιστούμε στον κανονισμό 78, για παράδειγμα, για την προστασία των πεζών. Ό,τι ισχύει δηλαδή στις οδικές μεταφορές. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και εδώ όταν πρόκειται για το σχεδιασμό και τις δοκιμές ε, που γίνονται των υλικών για να ε, μειωθούν τα θύματα. Ξέρουμε, έχουμε υπόψη μας, διάφορες περιπτώσεις τραγικών ατυχημάτων, κολυμβητών. από τέτοια σκάφη. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την προσέγγιση που ισχύει για τους πεζούς. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε την ίδια προσέγγιση και εδώ όταν μιλάμε για τον σχεδιασμό τέτοιων σκαφών αναψυχής. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή για την συνεργασία του. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας με νέες προτάσεις και ίσως συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ρούβεξ είναι εδώ. Όχι. Κανένας άλλος που θέλει το λόγο, παρακαλώ, πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλώς, Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Κύριος Γκυράουλ, είσαστε εκεί. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ε, ευκαιρία να διευκρινίσουμε ορισμένα από τα ζητήματα που έθεσαν οι ευρωβουλευτές. Με κάθε σεβασμό λοιπόν τώρα στην έκθεση του κύριου Ζήλη και τα σχόλια που έγιναν. Εμείς θέλουμε να επενθυμίσουμε ότι έχουμε κάποιες δυσκολίες με το τελικό τμήμα των τροπολογιών 2 και 5 στην έκθεση του κυρίου Δήλη. Όσον αφορά τις νέες τροπολογίες, έχουμε δυσκολίες με πολλές από αυτές. Συνεπώς, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, 8 για παράδειγμα. Εμείς εδώ πέρα μιλάμε για τη λογική σκέψη, δεν μιλάμε για άρθρο. Τροπολογία 9. Δεν νομίζω ότι πρέπει να επεκταθεί η αιτιολογική σκέψη, γιατί μιλάμε για τους ορισμούς. και λαμβάνουμε υπόψη μας εδώ τις απαιτήσει και τη στήριξη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι στην τροπολογία 10. Εμείς πιστεύουμε ότι πρόκειται περισσότερο για ένα οριζόντιο ζήτημα, γιατί μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη πράξη πρέπει να χαίρουν ιδιαίτερη προσοχής. Τώρα τι ειδική στήριξη μπορεί να προβλεφθεί, εδώ υπάρχει ερωτηματικό δεν κωδικοποιείται. Για την τροπολογία 11. Εντάξει. Mm. Τροπολογία 12. Τη στηρίζουμε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπαίνει στις εμπορικές δραστηριότητες. Τροπολογία 13 και τροπολογία 20. Έτσι όπως τη διαβάζουμε εμείς, δίνει τη κατεξοδότηση εξουσίες στην Κομισιόν ενώ δεν το έχουμε ζητήσει και δεν πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να επεκταθούν οι αρμοδιότητες αυτές όσον αφορά τα επίπεδα εκπομπών. Τροπολογία 14. Καταρχήν δεν πιστεύουμε ότι χρειάζεται. Αλλά θα μπορούσαμε να δεχτούμε το τελευταίο τμήμα της τροπολογίας αυτής. Το ενδιάμεσο, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε εμείς, είναι υπερβολικό. Τροπολογία 15. Εντάξει, 16. Είμαστε ανοιχτοί στον ορισμό των υβριδικών, μάλλον συγγνώμη, των αμφίβιων σκαφών. Δεν νομίζουμε ότι είναι πρόβλημα αυτό. 17. Είναι περιττή. 18. Καλύπτεται ήδη από το άρθρο 5. Και επιπλέον έχει να κάνει με μια ειδική κατηγορία σκαφών. Δεν θα έπρεπε, πιστεύω εγώ, κάποιες κατηγορίες να απομονώνονται από τα μέτρα. Έρχομαι τώρα στην τροπολογία 19 έτσι όπως διατυπώνεται δεν είναι ορθή κατά τη γνώμη μας. Θα μπορούσαμε όμως να δεχτούμε τη δυνατότητα να επαναλάβουμε αυτά τα οποία υπάρχουν και στο άρθρο 22 πρώτη παράγραφος που αναφέρεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Τροπολογία 20. Σας είπα για αυτήν. 21. Πρόκειται για τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Είμαστε ανοιχτοί να συμπεριλάβουμε οτιδήποτε υπάρχει στην ε, διοργανική συμφωνία, οπότε αν πρέπει να αλλάξει κάτι στο κείμενο αυτό δεν είναι πρόβλημα για μας. Τροπολογία 22. Όπως είπε και ο κύριος Σίλια, εδώ πέρα υπάρχουν ε, απαιτήσει για την ε, προβολή, για το ορατό. Επιπλέον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε έναν ευρύ κατάλογο ατυχημάτων ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε τι προβλήματα θα μπορούσαμε να λύσουμε. Συνεπώς θα προτιμούσαμε να αφήσουμε το κείμενο ως έχει. Να μην συμπεριλάβουμε δηλαδή την προσθήκη αυτή που ζητάει η τροπολογία 22. Στην έκθεσή μας που θα έχει να κάνει με την εφαρμογή του μέτρου θα μπορούσαμε τότε να δούμε το θέμα αυτό της δηλαδή, αναφοράς των ατυχημάτων. Για την τροπολογία 23. Είπαν κάποια κράτη-μέλη ότι πρέπει να διευκρινιστεί η απέτηση αυτή. Γιατί δεν είναι σαφές το τι πρέπει να γίνει. Τι ζητά ακριβώ αυτή η τροπολογία. Και είναι επικίνδυνο βέβαια αν κάποιος πέσει από το σκάφος, ε, όντως δεν είναι εύκολο να επανέλθει. Θα μπορούσαμε λοιπόν ενδεχομένω να δεχτούμε την τροπολογία αυτή ως προστίκη στο τέλος δηλαδή του κειμένου που προτείνει η Επιτροπή μπορούμε να προσθέσουμε αυτό ότι θα υπάρχει ε, πρόσβαση ε, για κάποιον άνθρωπο που βρίσκεται αβοήθητο στο νερό. Τώρα, στη συνέχεια, πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποια παρεξήγηση εδώ σε σχέση με τόσα αναφέρει η έκθεση αντικτύπου. Γιατί? Γιατί αυτό το οποίο αναφέρεται εκεί, τεχνικά μιλώντας, είναι εφικτό να μειωθεί ο θόρυβος κάποιων κινητήρων. Αλλά μιλάμε για τον θόρυβο που προκαλείται από το σκάφος. υπάρχει η μείωση του επίπεδου θορύβου του κινητήρα, αλλά πρέπει να δούμε και συνολικά τους σκάφους. Τα περισσότερα προβλήματα τα έχουμε σήμερα από σκάφη, τα οποία απόλυτα νόμιμα κυκλοφορούν, αλλά έχουν ε, αρχίσει να κυκλοφορούν πριν μπουν οι προδιαγραφές για τον ήχο. Ενώ τώρα δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές αυτές. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μας, αν θέλουμε επιπλέον περιορισμό στην ηχορύπανση, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. <clears throat> Και επιπλέον αυτό σημαίνει νέο σχεδιασμό των σκαφών, προκειμένου αυτά να μπορούν να τα αποκριθούν στις νέες αυτές προδιαγραφές. Και ο επανασχεδιασμός αυτός, όπως καταλαβαίνετε, κοστίζει πάρα πολύ. Αυτά. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλες διευκρινήσεις θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ο Ζήλα. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους που πήραν το λόγο, τους σκιώδες εισηγητές για την ε, επικοδομητική συνεργασία πρώτα απ' όλα που είχαμε μεταξύ μας. Αλλά θέλω να αναφερθώ στις θέσεις των διαφόρων κομμάτων. Τροπολογία 9 από το ΑΛΚΑ. Η προφορική τροποποίηση δεν αλλάζει τίποτα. Είμαστε κατά της τροπολογίας 9 έτσι κι αλλιώς. Τροπολογία 10 Θα χρειαστεί κατά τμήματα ψηφοφορία, γιατί εμείς είμαστε σύμφωνοι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την στήριξή τους. Αλλά το τελευταίο που μιλάει για παρεκκλήσεις, εκεί δεν πιστεύουμε ότι είναι αυτό που θέλουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει για την τροπολογία 23 να προσθεθεί αυτό το οποίο ζητήθηκε από τους πράσινους. Ναι. Σχετικά με, το, με την πρόσβαση ατόμων ε, αβοήθητων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ζήλε. Θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί στις 9 και 10. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη τώρα. Έκθεση για τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Συνδρομικό Χώρο. Η συγγήτρια, η κυρία Σερακιάνη. Το Νοέμβριο τη ζητήθηκε να ξεκινήσει τριμερή διάλογο. Το Συμβούλιο ανέκρινε την θέση της στις 11 Μαρτίου. Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε στους συντονιστές η να ενημερώσει για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και σήμερα είναι ο πρώτος επίσημος τριμερής διάλογος με τη συμμετοχή της ε, μόνιμης αντιπροσωπείας της Δανίας εκ μέρους της Προεδρίας βέβαια. Ακριβώς πριν από τη δικιά μας συνεδρίαση έγινε η συνάντηση αυτή. Μην ξεχνάμε ότι στόχος μας είναι η δεύτερη ανάγνωση και η διαδικασία προβλέπει να εγκρίνει το Σεβούλιο την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου χωρίς τροποποίηση. Αυτό σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις ε, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δεύτερη ανάγνωση, πριν την Ολομέλεια του Ιουλίου, τη δικιά μας. Οπότε, πρέπει να τηρήσω την διαδικασία όπως καταλαβαίνετε και άρα τη δεύτερη ανάγνωση να την έχουμε ολοκληρώσει στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Κύριε Σαρακιάνη, έχετε το λόγο για να μας ενημερώσετε επί των διαπραγματεύσεων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και εσείς είπατε, από τον Ιανουάριο υπήρξαν άτυπες συναντήσεις με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Προφανώς η θέση του Συμβουλίου είναι πιο ήπια, ακόμη και σε σχέση με το κείμενο της Επιτροπής. Συμμερίζομαι τις ε, θέσεις της Επιτροπής όμως, όπου λέω ότι σε κάποια ουσιώδη σημεία της αναδιατύπωσης, η θέση του Συμβουλίου είναι υπερβολικά ήπια. Υπήρξαν επικοδομητικές συζητήσεις βέβαια σήμερα και επειδή σήμερα είχαμε τον πρώτο επίσημο τριμερή διάλογο, ακριβώς πριν τη συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής, εξετάσαμε 7 σημεία του διτακτικού που ήταν πολύ σημαντικά, 7 σημεία της αναδιατύπωσης και επειδή ο εξαρτών βρήκαμε ήδη ε, συμβαστικές λύσεις για τα 5 υπόλοιπα, τουλάχιστον για τα 3 νομίζω ότι θα μπορέσει με διαλλακτικότητα από την πλευρά όλων να βρεθεί κάποια συμφωνία. Βεβαίω, για κάποια σημαντικά σημεία ακόμη υπάρχουν ε, διαφωνίε. Για λόγου σαφήνεια, θα θέλω να παραμείνω στα πιο ουσιώδη σημεία τη αναδιατύπωση, ξεκινώντα από τον ε, ρυθμιστή, που είναι το καθοριστικό μέρος της σιδηροδρομικής αναδιατύπωσης, κάτι που συζητήσαμε και σήμερα, και έπειτα Υπάρχουν και τα θέματα που σχετίζονται με τη βούληση του Κοινοβουλίου να υπάρχει ανεξάρτητος εθνικός ρυθμιστής, ισχυρός, με πόρους στη διάθεσή του και τη δυνατότητα να εφαρμόσει κανόνες παρόμοιους, ίδιους, για τις 27 ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ η συζήτηση ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη, διότι το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση είχε θεωρήσει ότι τα εθνικά κοινοβούλια είναι εκείνα που πρέπει να διορίζουν τους ρυθμιστές. Ενώ το Συμβούλιο θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν εκτελεστικοί φορεί Η κυβέρνηση η Προεδρία του Συμβουλίου που να αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη. Νομίζουμε λοιπόν ότι στο σημείο αυτό η διαφωνία παραμένει, όμω ελπίζουμε ότι μια διατύπωση εν μέρη διαφορετική από αυτή που το Συμβούλιο μα υπέβαλε θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Κατά τα άλλα, για πολλά σημεία που αφορούν τους κανόνες του ρυθμιστή έχουμε ήδη συμφωνήσει και εργαζόμαστε για να βρούμε μια λύση ικανοποιητική εντός ε, προθεσμίας. Για την χρηματοδότηση. Που κατά κάποιο τρόπο προσπαθήσαμε να κάνουμε πιο σταθερή με την πρώτη μας ψηφοφορία σε ό,τι αφορά τις συνδροδρομικές υποδομές. Θεωρούμε εδώ ότι η συμφωνία που βρήκαμε για την πολιτική σύμβαση και τη διάρκεια τη είναι σημαντική. Υπήρχαν και εδώ διαφορετικές απόψεις. Το Κοινοβούλιο μιλούσε για τρία χρόνια. Το Συμβούλιο για επτά. Τελικά βρήκαμε τη μέση λύση των πέντε ετών. Και εδώ λοιπόν νομίζω ότι αποσαφηνίστηκε το θέμα αυτό και ήταν αρκετά σοβαρή επιτυχία. Βέβαια είναι προσωρινή όλη αυτή η συμφωνία γιατί μετά θα πρέπει να δούμε την ισορροπία τη συνολική του κειμένου. Αλλά επικοδομητική διάθεση υπάρχει από την πλευρά όλων ώστε να εξευρεθεί λύση. Όλοι οι συμμετέχοντες ε, έχουν τέτοια διάθεση. Σε ό,τι αφορά πιο συγκεκριμένα την ανεξαρτησία του διαχειριστή και την οικονομική διαφάνεια, συγκεκριμένα στο άρθρο 6, δεν προλάβαμε να εξετάσουμε το κείμενο. Θα θέλαμε εδώ να δούμε και κάποια πρόταση από την Προεδρία. Η μέθοδος που τώρα χρησιμοποιήσαμε ήταν παραγωγική ε, κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να ζητούμε πρόταση της ε, Προεδρίας και αφού υποβληθεί αυτή να τη χρησιμοποιούμε ως βάση για τη συζήτηση. Είναι ευαίσθητο το σημείο της χρηματοδότησης, αλλά έχουμε ακόμη περιθώριο για να διαπραγματευτούμε και καθώς βρισκόμαστε εν αναμονή της τοποθέτησης του Συμβουλίου, συζητήσαμε άλλα σοβαρά θέματα σήμερα. Τον θόρυβο, μετά από πρόταση της ομάδας των Πρασίνων, που υπέβαλε ο κύριος Κράμερ, κάτι που συμφωνεί με την θέση πολλών ε, βουλευτών και της Επιτροπής. Και εδώ ελπίζουμε ότι θα βρεθεί συμφωνία με το Συμβούλιο. Επίσης, όπως υπευλήθηκε η πρόταση για τα RTMS και τα GTS, CTS, και εδώ ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία, ακόμη και με τη δυνατότητα προσφυγής που θα αναλαμβάνει ο Εθνικός Ρυθμιστής. Το πρόβλημα δεν ήταν με τις κλασικές διαδικασίες, όπου αναγνωρίσαμε το δικαίωμα συμμετοχή όλων των μερών και με διάρκεια 6 εβδομάδων. Το θέμα είναι τι γίνεται με την περίπτωση όπου ο ρυθμιστής σε 30 ημέρε ζητά περισσότερα δικαιολογητικά, σχετικά έγγραφα δηλαδή, τεκμηρίωσης. Εκεί δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για την προθεσμία εντό τη οποία θα πρέπει να παραδοθούν τα έγγραφα. Δεν θέλουμε η διαδικασία τη προσφυγή να παραταθεί περιτά. Περιμένουμε λοιπόν εδώ ακριβώς την απάντηση του Συμβουλίου. Σε ό,τι αφορά τις βασικές ε, λειτουργίες του διαχειριστή της υποδομής και αυτό είναι καθοριστικό μέρος της αναδιατύπωσης και έχουμε ορίσει κάποια από τα βασικά καθήκοντα του διαχειριστή της υποδομής όπως η ανάρτηση, η παρουσίαση των δικαιωμάτων, η σήμανση αλλά και για την πρόσβαση στις υδροδρομικές υπηρεσίες. Μόλις σήμερα το συζητήσαμε και αυτό και στην ουσία συμφωνούμε στο μεγαλύτερο μέρος της πρότασης ε, όπως έχει υποβληθεί από το Συμβούλιο για το άρθρο 13 και το παράρτημα 2 αλλά δεν υπάρχει συμφωνία γιατί το Κοινοβούλιο ανέκαθεν θεωρούσε ουσιώδους σημασία την συντήρηση σε όλο αυτό το κεφάλαιο στο κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο αποκλείεται η συντήρηση ακριβώ. Εμεί αντιθέτω θέλουμε μεταξύ των βασικών καθηκόντων να περιλαμβάνεται η συντήρηση. Γι' αυτό συζητούμε ακόμα με το Συμβούλιο κατά πόσον μπορεί να γίνει μια αλλαγή που μα πρότεινε στο διτακτικό. Το Συμβούλιο, αλλά που εμεί ακόμη δεν έχουμε αποδεχτεί. Στην πρώτη ανάγνωση ζητήθηκε εξαίρεση για το, στην αναδιατύπωση με την συντήρηση για τις περιπτώσεις υψηλής ταχύτητας, όμως το Συμβούλιο κάνει μια διάκριση μεταξύ ελαφράς και βαριάς συντήρησης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον ε, μπορούμε να επιμείνουμε στο αρχικό κείμενο του Κοινοβουλίου. Εμείς δεν συμφωνούμε για την ώρα με τη δική τους πρόταση. Επίσης, το Συμβούλιο θέλει τη θέση σε ισχύ της νέας οδηγίας να την ε, μεταθέσει για 36 σε μερικά μέρη του κειμένου μήνες και για 60 σε κάποια άλλη. Εμείς επιμένουμε σε 12 μήνες για τη μεταφορά της οδηγίας, διότι θεωρούμε ότι ήδη έχει χαθεί πολύς πολύτιμος χρόνος. Οπότε θα πρέπει να εκινηθεί η διαδικασία σύντομα. Πρέπει αυτή η οδηγία να πάρει το δρόμο της με τρόπο αποτελεσματικότερο. Το άλλο ζήτημα που έχει και πολιτικό χαρακτήρα και ακόμη δεν έχει επιληθεί, το άρθρο 7, εκεί, μιλάμε για το άρθρο, που και το Κοινοβούλιο θέλει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άνοιγμα και διαχωρισμό των εθνικών αγορών το 2012 και 2013. Εδώ το Συμβούλιο έκανε πάλι μια πρόταση πολύπια. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε ακριβώς την διατύπωση λέξη προς λέξη. Αυτό συζητήσαμε σήμερα στην, στον τριμερή διάλογο. Ορίσαμε τώρα τις ημερομηνίε για τις επόμενες συναντήσεις, ε, των τριμερών διαλόγων δηλαδή. 9 Μαΐου και ακολούθως θα είμαι στη διάθεση των συναδέλφων βεβαίως για οποιαδήποτε διευκρίνηση και θέλω να ευχαριστήσω τους κοιόδους εισηγητές όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων για το έργο τους. Ήταν ε, πολύ δύσκολη δουλειά μας, αλλά νομίζω ότι υπήρξαμε παραγωγική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος μας κύριο Κούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κούν είναι στην Επιτροπή Αλίας, έχει άλλη έκθεση εκεί να παρουσιάσει. Οπότε εγώ θα παρουσιάσω τη θέση του ΕΛ και Ευχαριστούμε την εισηγήτρια για τη δουλειά των τελευταίων εβδομάδων. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες μόνο να υπενθυμίσω πως είναι σημαντικό για εμάς αυτή τη στιγμή να συνεχίσουμε να θεωρούμε ως σημείο κλειδί τις αρχές, τις ρυθμιστικές και με ειδικά τρεις πτυχές. Πρώτον, να είναι η αρχή αυτή ανεξάρτητη, να μπορεί να εργάζεται με τρόπο διαφανή και να έχει τα σχετικά μέσα. Δεύτερον, σταδιακά να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με τις εθνικέ διεθνιστικέ αρχές και τρίτον, η προθεσμία εφαρμογή να μην διαρκέσει μια αιωνιότητα και μια μέρα. Οπότε πρέπει να προβλέψουμε μια λογική προθεσμία. Αν επιτύχουμε αυτά τα πράγματα και αν θυμηθώ την ψηφοφορία, Νομίζω πως μπορώ να πω πως θα έχουμε στείλει ένα πολύ θετικό μήνυμα και βεβαίως ε, έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε και στο unbundling ε, γιατί βεβαίως ένας, ε, μια ισχυρή ρυθμιστική αρχή μπορεί να παίξει θετικό ρόλο. Χαιρόμαστε για κάποιους συμβιβασμούς που ευρέθησαν σήμερα, δηλαδή τις τελευταίες μέρες, ειδικά τα πέντε έτη για το κόστος των υποδομών και εγώ διαπίστωσα πως το Συμβούλιο συχνά είναι υπέρ μιας ε, εξαίρεσης για τη Βαλτική. Εγώ είμαι πεπισμένος πως σε άλλα σημεία θα πρέπει να ε, καταφέρουμε κάποια πράγματα. Τώρα αν μιλάμε για τις ουσιαστικές υπηρεσίες ή το άρθρο 7... Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να είναι ξεκάθαρο προς τα έξω. Στην συζήτηση περιοριστήκαμε στη ρυθμιστική αρχή με την υπόσχεση πως η Κομισιόν σύντομα, δηλαδή 2012, αλλά από ό,τι φαίνεται μπορεί να είναι και αρχές του 2013, να κάνει προτάσεις για το unbundling, για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό. Και ανεξαρτήτως ε, του ποια είναι διατύπωση, σημαντικό για μένα είναι τι έχει πει η Κομισιόν. Θεωρώ πως αυτό είναι μέρος της δικαιοσύνης εδώ πέρα στην Επιτροπή. Κάποιοι συνάδελφοι δεν έθεσαν ορισμένα ζητήματα και είναι και θέμα δικαιοσύνης στις διαπραγματεύσεις. Οπότε υποθέτω πως είναι σημαντική αυτή η ε, διατύπωση. Τώρα γρήγορη λύση θα είναι βεβαίως και έγκαιρη θα είναι θετική γιατί όλα αυτά τα οποία λέμε έχουν νόημα μόνο εάν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει με αυτό το πακέτο. Δεν θα ήταν σωστό να συζητάμε το επόμενο πακέτο πριν ολοκληρώσουμε το τωρινό. Αυτά και ευχαριστώ την Κομισιόν και τους ε, εκπροσώπους του Κοινοβουλίου που έκαναν καλή δουλειά. Ευχαριστώ κυρία Τρεμόζα. Εγώ, εγώ είμαι ο κύριος Τρεμόζα σήμερα. Μάλιστα. Όλα, όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Και δεν θα μιλήσω ισπανικά όμως. Θα μπορούσα, θα μπορούσα αλλά δεν το κάνω. Θέλετε να μ' ακούσετε τώρα τι θα πει η Άλντε. Ναι, λοιπόν, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον εισηγητή. Ο κύριος Τρεμόζα δυστυχώς δεν μπορεί να παραβρεθεί σήμερα. Οπότε θα τα εγώ που είμαι η ε, συντονίστρια, με συγχωρείτε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι κάποια πράγματα θετικά. Θα ξεκινήσω από τα μικρά και θα έρθω στα μεγάλα. Παραδείγματο χάρη. Από τη σκοπιά του εισηγητή μα του κυρίου Τρεμόζα, είναι σημαντικό η Κομισιό να μην έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο. Σημαντικό είναι για μας να υπάρχει ένας χρόνος για την εφαρμογή που θα είναι τουλάχιστον 12 μήνε. Όσον αφορά τη συντήρηση, αυτά τα οποία μας είπε η κυρία Σερακιάνη, που θέλει να τα βγάλει αυτά έξω το Συμβούλιο. Κοιτάξτε, κατά την απόψή μα ε, μετά από αυτά τα οποία ακούσαμε, ε, νομίζω λογικό είναι μακροπρόθεσμα να συμπεριληφθεί και η ε, συντήρηση. Εντάξει, μπορεί να προσπαθεί να τα κρατήσει εκτός το Συμβούλιο, αλλά είχαμε διαφορετικές ε, πληροφορίες από τους γερμανικού σιδηρόδρομους. Ξέρετε, τα πράγματα δεν είναι παντού συμβατά και είναι κρίμα αυτές οι δύο μεγάλες ε, σιδηροδρομικές εταιρείε που αναφέρθηκαν προσπαθούν ε, και να μην μπορούν να βελτιώσουν την συμβατότητα. Α δούμε τι μπορεί και τι πρέπει να βελτιωθεί. Τώρα για το ε, ρεύμα και την τιμή του το ρεύμα το σιδηροδρομικό. Εμείς είμαστε πάντα υπέρ της διαφάνειας ε, στον ανταγωνισμό. Και τέλος τα δύο σημαντικότερα πράγματα για εμάς είναι σημαντικό να μην χάσουμε το στόχο της ιδιοκτησιακής αποδέσμευσης και διαχωρισμού ε, αναρωτιόμαστε, η Κομισιόν ε, θα καταθέσει φέτος ε, πρόταση. Είχαμε πει πως δεν είναι αυτό το βασικό βεβαίω, το βασικό είναι η ισχυρή ρυθμιστική αρχή, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός. Και μας ενδιαφέρει το εάν θα υπάρξει και διαχωρισμός και διαφάνεια στα, στις χρηματικές ροές, έτσι ώστε το κόστος να ρέει ξανά στην ε, υποδομή για, ένα, για μια μίνι, ένα διαχωρισμό. Και βεβαίως χρειάζεται και ισχυρός εθνικός και ευρωπαϊκός ρυθμιστής. Ξέρω πως εδώ πέρα δεν συμφωνούν οπωσδήποτε όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες, οπότε εδώ πέρα χαίρομαι για αυτά τα οποία λέει η κυρία Σερακιάνη. Και ελπίζω να μπορέσουμε στο τέλος να συμφωνήσουμε και να υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κράμερ για τους πράσινους. Θα επαναλάβω τα όσα ακούστηκαν. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές. Δεν είναι απλό να βρει μια θέση. Ήδη στις προκαταρκτικές συζητήσεις θα ήθελα να αφαιρθώ σε τρία πράγματα. Έχουμε το θέμα του θορύβου και το θέμα ERTMS εντύπωσή μας ήταν πως ε, το Συμβούλιο το είχε καταλάβει, έτσι μας είπαν, αλλά βεβαίως μηδένα απρό του τέλους μακάριζε. Θα δούμε τι θα μου γίνει στην ουσία. Βεβαίω, ε, το βασικό θέμα είναι η ρυθμιστική αρχή. Ε, σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς στο Κοινοβούλιο. Θα είναι σκληρή η αντιπαράθεση οπωσδήποτε και μετά όταν ξεκαθαρίσουν όλες τις θέσεις, πότε θα τεθεί εν ισχύ. Και ο Ματιέ, ξέρεις, ανάμεσα στο χτες και την αιωνιότητα ε, μεσολαβεί μεγάλο διάστημα. Γι' αυτό εμείς ε, επιμένουμε στις 12 μήνες ή το σύντομο διάστημα, γιατί πάντα λέμε πως ε, έχουν περάσει ήδη 60 μήνες. Αν περιμένουμε άλλα 5 χρόνια, τι θα γίνει εδώ πέρα. Δεν, δε γίνει νόμοι αυτοί. Οπότε αν παραμείνουμε ενωμένοι νομίζω πως θα μπορέσουμε να περάσουμε και μια ισχυρή ρυθμιστική αρχή που θα είναι ανεξάρτητη. Εδώ πέρα συμφωνούμε όλοι. Πρέπει να δούμε βέβαια λεπτομέρειες, να προσέξουμε και το πως θα διασφαλιστεί η ανεξαρτησία. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει και εδώ πέρα μία ε, προθεσμία, όχι να μας λένε δεν συμπληρώθηκαν τα έγγραφα και να το χρησιμοποιούν για παραθυράκι να περάσουν 2-3 χρόνια. Όχι. Πρέπει να υπάρξει μια προθεσμία. Το πολύ δε ε, μετά από 8 εβδομάδες ε, να υπάρχει αντίδραση, γιατί αν ενδιαφέρονται και οι δύο πλευρές για την κρίση της υποδομής και λείπει κάτι, τι γίνεται, έρχονται σε επικοινωνία, σε τρει μέρε ξέρουν τι λείπει. Ε, δηλαδή, αν θένε να το κάνουν, γίνεται τσακ, τσακ, τσακα, Αλλά άμα δεν θένε, ξέρετε, λείπει η τάδε σφραγίδα και το τάδε έγγραφο και άμα θένε το τρενάρουν πάρα πολύ. Αλλά νομίζω πώς θα το περάσουμε αυτό. Αυτά τώρα θα τα δούμε τα υπόλοιπα στις ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριο Ζήλε. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια. Ναι, για να με παρακολουθήσετε χρειάζεστε βοήθεια. Λοιπόν, ευχαριστώ τους συναδέρφους, τους σκιώδεις εισηγητές. Θέλω όμως να αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Πρώτον, το Συμβούλιο συναντήθηκε σήμερα. Η συνδιαλλαγή ασχολήθηκε κυρίως με την ανεξαρτησία των εθνικών ε, ρυθμιστών και εδώ κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε αδιέξοδο. Αν επιμείνουμε στην εκδοχή της πρώτης ανάγνωσης που λέει ότι είναι τα εθνικά κοινοβούλια εκείνα τα οποία ορίζουν τους εθνικούς ρυθμιστές, τότε δεν δημιουργούμε περισσότερη ανεξαρτησία για τον ρυθμιστή αυτόν. Ο ρυθμιστής ήταν ένα διαμεσολαβητή κατά κάποιο τρόπο μεταξύ διαφόρων χωρών ε, μελών για την προσβασιμότητα στα δίκτυα. Ίσως λοιπόν οι εθνικοί ρυθμιστές να μην είναι αντικειμενικοί και να θέλουν να υποστηρίξουν τα συμφέροντα της δικιάς τους χώρας. Έχουμε 27 χώρες μέλη και η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Συνεπώς, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να πετύχει κανείς την ανεξαρτησία των ρυθμιστών. Αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ζητάω από τους συναδέλφους να το σκεφτούν. Το δεύτερο θέμα είναι το πώς θα ολοκληρώσει τη δουλειά του ο ρυθμιστής. Έξι μήνες προτείνει το Συμβούλιο. Έξι μήνες να μην μπορεί να δουλέψει σε καμία εταιρεία ο ρυθμιστής για την οποία να έχει πάρει κάποια απόφαση. Για μας η περίοδος αυτή πρέπει να είναι δύο χρόνια. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών, κάπου να είναι λίγοι μήνες και αλλού να είναι δύο χρόνια. Αυτό ισχύει σήμερα. Αλλά το πιο συνηθισμένο είναι δύο χρόνια και για μένα αυτό θα πρέπει να προτείνουμε. Κάτι ακόμα. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να μας στηρίξουν για το σημείο 17 όσον αφορά την προσβασιμότητα τρίτων ε, χωρών, δικτύων τρίτων χωρών. Κυρίως όταν πρόκειται για εμπορικές μεταφορές ε, μέσω σιδηροδρόμου. Στις βαλτικές χώρες, για παράδειγμα, έχουμε ανταγωνισμό ε, από ρώσικες εταιρείες. Αν δεν μας στηρίξετε σε αυτό, θα βρεθούμε σε μειονεκτική θέση, γιατί εμείς έχουμε ένα πιο φιλελεύθερο σύστημα. Αν δηλαδή επιτρέψουμε ένας μια ρωσική επιχείρηση να μπορεί να πηγαίνει από τη Μόσχα στο Βίλνιους, στη Ρήγα κτλ. Ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να δουλεύουν μόνο στο κομμάτι του δικτύου που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνετε ότι θα βρεθούμε σε σοβαρά μειονεκτική θέση. Θα πτωχεύσουν οι δικές μας οι επιχειρήσεις, η αξία τους θα μειωθεί κατά πολύ θα βγουν από τη μέση. Σας υπενθυμίζω ότι για πολλά χρόνια στις βαλτικές ε, χώρες ήμασταν ε, και αγωνιστήκαμε κατά των διακρίσεων στις τιμές. Αν κάποιος τώρα μεταφέρει εμπορεύματα από την Μόσχα στο Αγίο Πετρούπολη έχει μία τιμή. Αν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάει στη Ρήγα ή αλλού πρέπει να πληρώσει πολύ περισσότερα. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν μιλάμε για το άνοιγμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου σε τρίτες χώρες. Δεν πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά ελαφρά την καρδία. Μην κάνουμε γεωπολιτικά σφάλματα. Ζητάω από του συναδέλφου να τα σκεφτούν όλα αυτά πολύ σοβαρά. Φυσικά και μπορεί να υπάρχουν κάποια νομικά εμπόδια, όπω είπε σήμερα η Επιτροπή στη συνάντηση. Είμαι όμω πεπισμένο ότι πρέπει να βρούμε μία διέξοδο. Το έχουμε κάνει και άλλη φορά. Τέλο, ξέρετε ότι εγκρίναμε την οδηγία για το φυσικό αέριο το 2009. Αυτό σημαίνει ότι οι υποδομές φυσικού αερίου είναι τέτοιες ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι. Οι τρίτες χώρες είναι κατά της εφαρμογής των ε, κανόνων αυτών πλήρους και η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα δεν μπορεί να πιέσει επ' αυτού τις τρίτες χώρες. Μα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό στον εαυτό μας και να υποστηρίζουμε τα δικά μας τα συμφέροντα όταν πρόκειται για τέτοια νομικά κείμενα όπως είναι αυτό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, στα πλαίσια του τριμερούς αυτού διαλόγου που γίνεται με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, θέλω να επαναλάβω ότι η τροπολογία 135 που έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τεράστια σημασία. Στηρίχθηκε στην Ολομέλεια από όλε τι πολιτικέ ομάδε με πάνω από 430 ψήφου υπέρ. Πρέπει να θυμόμαστε ότι σε ορισμένες χώρες μέλη έχουμε αυτοχρηματοδότηση στους σιδηροδρόμους, στους συνδρομικούς φορείς. Και δεν υπάρχει σύνδεση ούτε με τα εθνικά δίκτυα ούτε με τα ευρωπαϊκά. Για τους φορείς αυτούς λοιπόν, αν ε, θέλουμε να εφαρμόσουν όλες τις προδιαγραφές της οδηγίας, αυτό θα σήμαινε δυσανάλογο βάρος και θα ήταν κατά του πνεύματος της οδηγίας. Συνεπώς, θα έπρεπε να υιοθετήσουμε λύσεις οι οποίες να βοηθήσουν τις χώρες μας να αναπτυχθούν θετικά. Αλλιώς ρυθμίζουμε υπερβολικά την αγορά, κάτι το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε. Ο κύριος Ελκαντράουι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα βεβαίως να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική έκθεση, τη δουλειά που έχει κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περιοριστώ στο να τονίσω το ότι είναι σημαντικός διαπραγματεύσεις, το ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι, ο ρόλος δηλαδή της ε, ρυθμιστικής ε, αρχής. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Ποιο είναι δηλαδή το σημαντικότερο κατά την άποψή μας. Να είναι ισχυρός, ανεξάρτητος, να μπορεί να αντιδρά, να παρεμβαίνει και δεδομένου του ότι τα δίκτυα, οι ρυθμιστικές αρχές είναι εθνικές και οι γραμμές διεθνείς να δημιουργήσουν ένα δίκτυο ρυθμιστικών αρχών. Σημαντικό αυτό για τους χρήστες, ε, τους πελάτες, ε, για να μπορούν εύκολα να απευθυνθούν σε κάποιον ε, για τα προβλήματά τους. Ειδικά όσον αφορά τη λειτουργία της αγοράς που πρέπει να υπάρχει ενιαία ερμηνεία της παντού στην Ευρώπη. Βεβαίως, μακροπρόθεσμα, η ιδέα μιας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής, δεν έχουμε φτάσει εκεί, αλλά είναι κάτι στο οποίο πρέπει να κάνουμε τα πρώτα βήματα. Επίσης, θεωρώ πως μια ισχυρή ρυθμιστική αρχή είναι σημαντική όσον αφορά και τις χρηματικές ροές εντός μιας επιχείρησης σιδηροδρομικής και μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα για να μπορεί να κρίνει το εάν οι χρηματικές αυτές ροές ε, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και τη λειτουργία της αγοράς. Σε μια μεταγενέστερη βάση βέβαια θα γίνει μια πιο ουσιαστική συζήτηση το επόμενο έτος για την ε, αποδέσμευση την ε, ιδιοκτησιακή το unbundling που λέμε και αναμένουμε με αγωνία την πρόταση της Κομισιόν. Βεβαίως, πρέπει να δούμε τη λειτουργία της αγοράς και την αποτελεσματικότητα του σιδηροδρομικού δικτύου και το κόστος ε, που θα έχει ο διαχωρισμός. Αυτά. Δεν μπορώ. Συνέχισε έτσι. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μπάνια. Ε, yeah, yes, uh, forgive me for being... Με συγχωρείτε που δεν έχω μελετήσει προσεκτικά το έγγραφο αυτό. Απλώς διερωτώ με, η τροπολογία είναι για την εξαίρεση. Είναι η μόνη εξαίρεση που συζητήθηκε. Είναι προσθήκη σε άλλες προπάρχουσε εξαιρέσει. Διότι υπάρχουν σιδηροδρομικά δίκτυα αποκομμένα από το υπόλοιπο. Θα ξέρετε τι εννοώ, Δερεμή. Όταν συζητήσαμε την αποσύνδεση στο Ηνωμένο Βασίλειο στο διαχωρισμό. Ίσως να μην ήταν η καλύτερη δυνατή μέθοδος, αλλά κάτι καταφέραμε. Νομίζω ότι το αλικό δίκτυο λόγου χάρη πήρε μια τέτοια εξαίρεση για το βρετανικό σύστημα. Δηλαδή, το διαχωρισμός θα επιβληθεί σε όλα τα σιδηροδρομικά δίκτυα. Υπάρχουν και ιδιαίτερε καταστάσεις σιδηροδρομικά δίκτυα, τα οποία είναι τελείως αποκομμένα από το γενικότερο δίκτυο, που εξαιρούνται και για άλλους λόγους. Κύριε Μπάνιεν, τι εννοείται ακριβώ, οι συνάδελφοι δεν το καταλάβουν. Αυτοί οι ιστορικοί σιδηρόδρομοι εξαιρούνται για όλου του ε, δυνατού λόγου και όλοι γνωρίζουν γιατί έχουν εξαιρεθεί για την ίσο του White. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε για ιστορικό σιδηρόδρομο, αλλά τέτοιου, έχουμε κάποιες φορές που κάποιους τέτοια δίκτυα που λειτουργούν και σε διαφορετικές τροχές και ράγες και γι' αυτό και εξαιρούνται. Θα ζητήσουμε την Επιτροπή μια διευκρίνηση για τον ίσο του White αλλά το Ρωμανό Βασίλειο μπορείτε να μην το ζητά για καν αυτό που λέτε. Ο κύριος Καντζάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όσους εργάστηκαν για το θέμα αυτό και όσους το συντονίζουν βεβαίως. Την κυρία Σερακιάνη δηλαδή. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι ενδεχομένως να υπάρχει τρόπος να ξεπεράσουμε το μπλοκάρισμα που δημιουργήθηκε στην πρώτη ανάγνωση. Γι' αυτό και δεχτήκαμε να συμπεριληφθεί σε αιτιολογική σκέψη το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει πρόταση για την απελευθέρωση των εθνικών αγορών για επιβάτες αλλά και για τη διάρθρωση των εταιριών που λειτουργούν στην αγορά. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προχωρεί σε σχέση με αυτό μας το αίτημα πρόκειται να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που προβλεπόταν. Και πιο συγκεκριμένα νομίζω ότι έχουμε την υποχρέωση και το καθήκον να απελευθερωθούμε από φραγμούς και περιορισμούς, να καταστήσουμε ανταγωνιστική την αγορά. Εάν πράγματι θέλουμε να επιδιώξουμε το στόχο, το στόχο μας δημιουργίας δηλαδή ενιαίου σιδηροδρομικού ευρωπαϊκού χώρου, θα πρέπει να τηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο τις φιλοδοξίες μας. Είναι ιδιαίτερη χρονική στιγμή. Ε, και αυτά τα χρονικά περιθώρια που έχουμε προβλέψει δεν συμπίπτουν με όσα μας ζητούνται εκτός Κοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να επιδείξουν όλη την καλή θέληση οι συνάδελφοι ώστε να προχωρήσουμε στην απελευθέρωση, στην άρση των φραγμών και να δημιουργήσουμε μια αγορά που να μας δώσει αποτελέσματα χειροπιαστά. Αυτό μας το ζητούν επισταμένως, δραματικά σχεδόν, οι πολίτες μας. Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος, διότι πολλά ήδη έχουν αναφερθεί. Θέλω να ενθαρρύνω την εισηγητριά μας, την κυρία Σερακιάνη, για ένα μακρόπνο εγχείρημα. Και το πρώτο που έχω να πω κάτι που πολλοί συνάδελφοι το ανέφεραν, είναι ότι στο άρθρο 7, εδάφιο 3, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μιλάμε εδώ για το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει οδηγία για την απελευθέρωση και την αποσύνδεση, το διαχωρισμό. Αυτό δεν ήταν απλώς ένα άρθρο. Αυτή ήταν η βάση για να εξευρεθούν ε, και άλλες συμβαστικές λύσεις. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα άκρος σημαντικό διότι η αναδιατύπωση τέθηκε σε αυτά τα θεμέλια ακριβώς. Υπήρξαν εδώ και ένα χρόνο κάποιες συγκεκριμένε υποσχέσεις. Να επιληφθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή αυτών των ε, θεμάτων και αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει καθορίσει την πορεία της για το θέμα αυτό. Και δεύτερη παρατήρηση σε σχέση με την ρύθμιση. Νομίζω όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για το ρυθμιστή, αλλά όπως είπε και ο κύριος Ελκαντάουι, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον ο ρυθμιστής θα είναι ρυθμιστής συνολικά εφόσον δημιουργηθεί ένας ενιαίο σιδηροδρομικό χώρο στην Ευρώπη και θέλουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των τρένων στην Ήπειρό μα. Ευχαριστούμε πολύ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Πάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σα. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντα την εισηγήτρια και του πιο εισηγητέ. Αλλά και η Προεδρία και όλοι μου οι συνάδελφοι έχουν εργαστεί εντατικά για το θέμα αυτό τι τελευταίε εβδομάδε και πριν τις κατά τις άτυπες συναντήσεις ε, να ετοιμάσουν συμβαστικές λύσεις. Είδαμε ότι δύο εγκρίθηκαν ε, στη σημερινή επίσημη συνάντηση του τριμερού διαλόγου. Δύο από τις εφτά λοιπόν προτάσεις έχουν καλυφθεί. Οι προσπάθειές μας λοιπόν ευωδόθηκαν και αυτό πραγματικά χαράζει τον δρόμο για να καταλήξουμε σε συμφωνία ε, στη δεύτερη ανάγνωση μέχρι το καλοκαίρι τουλάχιστον και αυτό επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό παρέχει όλα τη στήριξή τη και στην εισηγήτρια και στη συγκεκριμένη Επιτροπή και στην Προεδρία που, όπω ξέρετε, εργάζεται σε δυσχερεί συνθήκε. Με κοινή θέση στο Συμβούλιο που δεν ήταν εύκολο να εξευρεθεί πριν από λίγο καιρό. Βεβαίω κάποιε μετατροπέ θα πρέπει να επέλθουν στη θέση αυτή. Δεν ήταν απλό για την Προεδρία βεβαίω, αλλά έχει αναλάβει κάθε δέσμευση για να το πετύχει αυτό η Προεδρία. Είναι πάμπολε οι τροπολογίε, Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τι σχολιάσω όλε. Όμω προτείνω η Γραμματεία να εξετάσει τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι τροπολογίε αυτέ. Να πω ότι εγώ διακρίνω κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, γενικότερα κεφάλαια και ευχαριστώ την εισηγήτρια που πολλές φορές που πολλές φορές χρησιμοποίησε το κείμενο που είχε συμφωνήσει με την Προεδρία τη περασμένη εβδομάδα, όπω για τη Συμβατική Συμφωνία ή την πρόσβαση στι ρυθμισμένε υπηρεσίε ή την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην, ε, με, στην μεταφορά εμπορευμάτων με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Ήδη στην πρώτη ανάγνωση λοιπόν έχουμε εκφράσει τη συμφωνία μας για πολλά ζητήματα, αλλά η Προεδρία δεν έχει απαντήσει ή υποβάλει προτάσεις για πολλά άλλα. Εκεί λοιπόν θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε συμβεστικέ λύσεις, όπως για την εξαίρεση του χρονοδιαγράμματος που συζητήσαμε σήμερα, όμως εκεί δεν έχουμε ακόμη συμφωνήσει, ή για τις δαπάνες ITMS. Ξέρετε ότι αυτό το, υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε βελτίωση προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι πρόσδεκτη. Γι' αυτό το σύνολο τροπολογιών, απλώς όπως και η κυρία Σερακιάνη, να σημειώσω για την παρακολούθηση της συντροδομικής αγοράς ή της ρήτρας εκμίσθωσης υπήρξε πολύ θετική πρόοδος στην πρώτη μας συνάντηση σήμερα. Σε άλλες περιπτώσεις η συγγήτρια προτείνει να επανεισαχθούν τροπολογίες της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωκοινοβουλίου. Και στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις κάποια συμβαστικά κείμενα Εγκρίθηκαν από όλε τι πλευρέ, όμως για το σύνολο τροπολογιών εδώ, όπω και οι συγκεκριτές και οι συγκεκριτές τα γνωρίζουν, εμεί προτιμούμε τα συμβαστικά κείμενα αυτά όπω για τι προθεσμίες αποφάσεων των ρυθμιστών, της, ε, την πρόσβαση στι ιδροδομικές υπηρεσίε, την συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ομάδα την Ένωση των Ρυθμιστών. Όμω για το θέμα αυτό γενικότερα υπήρξε πρόοδο σήμερα. Επίση Πρόεδρε, υπάρχουν κάποιε τροπολογίε όπου στην πρώτη ανάγνωση ήδη είχαμε σημειώσει ότι ήταν δύσκολο να υπάρξει στήριξη, σε σχέση με τη δική μας τουλάχιστον αρχική πρόταση και τις μελλοντικέ μας υποθέσεις. Αυτό αφορά κυρίως τις 3, 8, 9, 11 και 14 που αφορούν την αποσύνδεση ή διαχωρισμό και εδώ θεωρούμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα έρθει προς τα τέλη της χρονιάς και αυτό θα σας επιβεβαιώσω ότι και για τα τρία ζητήματα, τρει δέσμε μέτρων ε, εργαζόμαστε εντατικά. Εδώ λοιπόν θα υπάρξει και σχετική αποτίμηση και πολλέ ανταλλαγέ μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων και συμμετεχόντων των τομέα και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βεβαίω που ετοιμάζουν αυτέ τι προτάσει. Στρατηγικό, λοιπόν στόχο ο Δεκέμβριο, το προσωπικό Τη γενική μα διεύθυνση ε, Μεταφορών αλλά και όσων εργάζονται για τι συνδρομικέ υπηρεσίες και δίκτυα εργαζόνται σκληρά. Παντώ σε σχέση με το διαχωρισμό, το unbundling, Τι τροπολογίε αυτές καλό θα ήταν να μην τις εγκρίνουμε έχουν, αλλά να δούμε τη γενικότερη ρήτρα που συζητιέται μεταξύ συγκεκριτρίας και προεδρίας και να καλυφθούν κατά αυτόν τον τρόπο για τα βασικότερα σημεία του διαχωρισμού και των ρυθμιστών, Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι ρήτρε αναθεώρηση και από τι δύο πλευρέ δεν είναι βέβαια ταυτόσιμε, αυτέ που προτείνονται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, όμω μπορεί να είναι σταθερά θεμέλια για να βρεθεί πολιτικός, λύση πολιτικού συμβέρου μεταξύ των δύο θεσμικών οργανών. Οπότε τελικά θα βρούμε κάποιο πεδίο συνεννόηση, ελπίζω, και για τα δύο θέματα αυτά. Σα ευχαριστώ ιδιαίτερω. Ευχαριστούμε, κύριε Πακέη την ίσως του White ξέρετε ή όχι. Κοιτάξτε, δεν το ξέρω, αλλά θα ρωτήσω. Ευχαριστούμε. Προθεσμία για την υποπολή τροπολογιών 33 μάλλον Μαΐου. Ψηφίζουμε στην Επιτροπή 31 Μαΐου. Στην Ολομέλεια του Ιουλίου θα περάσει το θέμα αυτό. Κύριε Σερακιάνη, θέλετε κάτι να προσθέσετε. Μόνο μια διευκρίνηση για τον Εθνικό Ρυθμιστή διότι ακριβώ ήθελα να διαφωτίσω του συναδέλφου. Ίσως το ξέχασα στην αρχική μου εισήγηση. Το Συμβούλιο στην αρχή δεν ήθελε καν να χρησιμοποιηθεί ο network, δίκτυο, δίκτυο δηλαδή ρυθμιστών. Εδώ έγιναν κάποια θετικά βήματα ω προ το θέμα του ρυθμιστή γενικότερα, οπότε συμπεριλήφθηκε αυτό το δίκτυο. Εδώ λοιπόν ευχόμαστε να υπάρξει το ενδεχόμενο να υπάρξει Ευρωπαίος ρυθμιστή. Αυτό επιδιώκουμε. Και σε ό,τι αφορά το άρθρο 7, επαναλαμβάνω, εμένουμε στι αρχικέ μα θέσει. Και για τον επιπλέον λόγο, τη διατύπωση που μα υπέβαλε το Συμβούλιο δεν θεωρούμε ότι είναι επαρκή. Όμως νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση που να κατευθύνεται προ την σαφήνεια που επιθυμούμε και τελικά όντω να υποβάλει και πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλο τη χρονιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σερακιάνη. Αν όλα πάνε καλά, οι διαπραγματεύσει θα συνεχιστούν ομαλώ και θα αποδώσουν και καρπού. Επόμενο σημείο στην εμερήσια διάταξη. Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Συζήτηση των τροπολογιών του κυρίου Ντεγκράντε Πασκουάλ. Η γνωμοδότηση. Κύριε Ντεγκράντε Πασκουάλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε το έτοιμά μου να ψηφίσουμε όχι αύριο, αλλά 7 Μαΐου. Και σας ευχαριστώ γιατί από την συνάντηση που είχαμε καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε λίγο χρόνο παραπάνω για να συζητήσουμε και να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε όσο γίνεται περισσότερο, περίπου σε όλα. Ακόμα δηλαδή και εκεί που δεν έχουμε συμφωνήσει μέχρι τώρα. ώστε να ψηφίσουμε και να συμφωνήσουμε όλοι. Κύριε Λουίς Δεγράντες, ε, μια στιγμή. Προηγουμένως να πω ότι όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν, να αποχωρήσουν ησύχως όμως. Χωρίς θόρυβο και φασαρία, αν μη τι άλλο δείξτε σεβασμό στον εισηγητή. Και συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά είχε πολύ φασαρία και δεν μπορούσαμε να σας ακούσουμε καλά. Ο εισηγητής, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έλεγα λοιπόν ότι η αναβολή θα χρησιμεύσει για να συνεχιστεί ο διάλογος ε, με τους σκιώδεις εισηγητές, διάλογος που είναι αναγκαίος. Έτσι κι αλλιώς ε, πάντα θέλω να έχω διάλογο με όσους υποβάλλουν τροπολογίες για να πετύχουμε συμφωνία, αν όχι πλήρη, αν μη τι άλλο, να περιοριστούν όσο γίνεται περισσότερο οι διαφορές μας. Ε, προτείνω πέντε συμβιβαστικές λύσεις ε, υπάρχουν και άλλες δύο που υπευλήθησαν. Συνεπώς, με όλες αυτές τις προτάσεις και δεδομένου ότι εγώ ως εισηγητής θέλω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όσο γίνεται περισσότερο, ε, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα σημεία στα οποία θα υπάρχουν διαφωνίες. Έτσι κι αλλιώς ένα είναι το σημείο στο οποίο διαφωνούμε. Είναι οι περίφημες 8 ώρες. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα πρέπει να ψηφίσουμε. Αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε και σε αυτό, δημοκρατικά θα ψηφίσουμε. Τι να κάνουμε. Θέλω όμως να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις, παρακαλώ, για το σημείο αυτό, για να εξηγήσω που ακριβώς διαφωνούμε. Σήμερα η Επιτροπή στατιστικά στα, στην Επιτροπή Γεωργίας θα εξηγήσει γιατί υπάρχουν οι διαφορές αυτές και γιατί δεν μπορούν να λυθούν. Πρέπει να ξέρουμε τα εξή. Ότι σχεδόν ποτέ δεν φτάνουμε στις 8 ώρες και ότι πρόκειται μόνο για ένα 37% των ταξιδιών, της μεταφοράς δηλαδή που γίνεται πάνω από 8 ώρες. Αυτό αναφέρεται στα στατιστικά στοιχεία. Επίσης, μόνο 40% των ζώων που μεταφέρονται πηγαίνουν για σφαγή. Και 60% είναι για πάχυνση. Και δεν καλύπτονται από τις τροπολογίες, μια που οι τροπολογίες αναφέρονται μόνο στα ζώα που πάνε για σφαγή. Τις προάλλες μπορέσαμε και συζητήσαμε και είπαμε ότι αν θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει συνοχή. Άλλο θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση στο ζώο που πηγαίνει για σφαγή από εκείνο το οποίο πηγαίνει για πάχυνση. Εδώ. Δεν έχω πρόβλημα να σας πω. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Διαπίστωση κάνω. Ότι πέρα από το θέμα της προστασίας των ζώων, τις άνεσής τους. Όλοι το θέλουμε. Κανένας δεν το αρνείται αυτό. Υπάρχουν συγκρόμενα συμφέροντα. Και μη σας εκπλήσει αυτό στην Επιτροπή Μεταφορών επίσης. Υπάρχουν χώρες οι οποίες ε, έχουν συμφέρον να πουλούν ε, κατεψυγμένα, άλλες ε, ζώντα ζώα, αλλού γίνεται η πάχυνση των ζώων είναι διαφορετική κατάσταση. Η Ολλανδία αγοράζει πολλά ζώα, πάνε στην Ισπανία κτλ. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε. Και για να σας εξηγήσω πληρέστερα για τους χείρους. 20 εκατομμύρια προέρχονται από τη Δανία και από την Ολλανδία, το 67% δηλαδή. Οι εξαγωγές των χώρων αυτών είναι για πάχυνση σε άλλες χώρες. Δηλαδή, αν συμφωνήσουμε με την γραπτή δήλωση, τα ζώα αυτά που ταξιδεύουν δεν θα συμπεριληφθούν. Γιατί στην ρύθμιση πρόκειται μόνο για ζώα τα οποία πηγαίνουν για σφαγή και όχι για πάχυνση. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα το οποίο μας διχάζει. Καλό θα ήταν όμως να είμαστε ειλικρινεί. Και θα ήταν καλό να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Και η Επιτροπή Γεωργίας προσπαθεί να καταλήξει σε συμβιβασμούς. Εγώ, Πρόεδρε, αν μη τι άλλο, και δεν θέλω εδώ να κάνω καμιά μιλία για να διχαστούμε ακόμα περισσότερο, απλώς να σας πω ότι υπάρχουν 40 τροπολογίες, οι 20 με αυτές με βρίσκουν σύμφωνο. Απλώς να σας εξηγήσω γιατί υπάρχει η κατάσταση που υπάρχει μεταξύ των σχεδόν εισηγητών. Νομίζω ότι το κλίμα είναι καρποφόρο και ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε περίπου σε όλα, εκτός από το περίφημο εκείνο των 8 ωρών. Είναι μια διαπίστωση, δεν θα συμφωνήσουμε. Τι να κάνουμε. Αν δεν βρούμε κάποια λύση με την οποία να συμφωνούμε όλοι, θα πρέπει να ψηφίσουμε και με δημοκρατικές διαδικασίες θα καταλήξουμε. Επαναλαμβάνω πάντως ότι είμαι υπέρ της προστασίας των ζώων, ότι διαπιστώνω πως η ρύθμιση της Επιτροπής έχει βοηθήσει πολύ και έχουμε πάει προς αυτή την κατεύθυνση ότι επιδέχεται βέβαια ο δρόμος αυτός ακόμα βελτιώσεις και συμφωνώ με την Επιτροπή για το ότι αυτό που χρειάζεται πάνω απ' όλα είναι η καλή εφαρμογή των κανόνων που ήδη ισχύουν. Αν δηλαδή ο κανονισμός εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο από όλου, είμαστε ήδη σε καλό δρόμο. Εν πάση περιπτώσει, Πρόεδρε, πρέπει να συζητήσουμε κι άλλο και ευχαριστώ που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε και να ξέρετε ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να συμφωνήσουμε περίπου σε όλα, Πρόεδρε. 7 Μαΐου λοιπόν παρακαλώ να ψηφίσουμε, όχι ακόμα για να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε. Τότε να ψηφίσουμε δημοκρατικά και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Έτσι θα λυθούν οι διαφορές μας. Επί της ουσίας αρμόδια είναι η Επιτροπή Γεωργίας. Από ό,τι φαίνεται και εκείνοι καταλήγουν σε κάποια συμφωνία. Θα μπορέσουν να το λύσουν. Δεν πρέπει να είναι ακαθόδες. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει την ευαισθησία των Ευρωπαίων πολιτών. Οπότε καλά κάνουμε εδώ και το συζητάμε. Με ειλικρίνεια και από την οπτική γωνία των μεταφορών, γιατί αυτό είναι ο ρόλος μας. Τίποτα άλλο, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Τεγκράντες. Ο κύριος Λάκφιτ, τη μέρου των Σοσιαλιστών, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σιγητά, σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα και για την ουσιαστική σας δουλειά. Θεωρώ πως σε πολλές προτάσεις που κάνατε είναι πάρα πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί δεν ε, απέχουν πάρα πολύ, αλλά θεωρώ πως για μένα και την ομάδα μου πως μπορώ να πω πως το ζήτημα των 8 ώρων ε, maximum διάρκειας ε, μεταφοράς είναι κάτι το ουσιώδες και θα κρίνει το εάν είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε με μια τέτοια έκθεση ή όχι. Θα ήθελα να προσπαθήσω να το εξηγήσω και ψυχρά, χωρίς συνέστημα. Βεβαίω, το θέμα είναι πως υπήρξε μια γραπτή δήλωση ε, που υπεγράφει από την πλειοψηφία των ε, βουλευτών. Και υπάρχει μια τάση της πλειοψηφίας, θα μπορούσε κανείς να πει. Αλλά το θέμα είναι πως εμείς ως αιρετοί εκπρόσωποι του λαού δεν μπορούμε να να μην ε, αντιδράσουν όταν ένας ΜΚΟ έχει συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν είναι μόνο αυτό σημαντικό. Επίσης υπάρχει λόγος για αυτές τις υπογραφές. Και δεν ασχολούνται έτσι για πλάκα αυτοί οι άνθρωποι να υπογράψουν. Υπάρχουν λόγοι. Οι λόγοι είναι δύο ειδών. Ε, ο πρώτος που είναι και για μένα πιο σημαντικός είναι ζητήματα αρχής, της προστασίας ε, των ζώων, ειδικά όταν μιλάμε για ζώα που πάνε για σφαγή ε, που θα πρέπει, που βεβαίως βλέπετε πως χειρίζονται διαφορετικά αυτά τα ζώα κάποια από ζώα τα οποία βεβαίως αξίζουν εκατομμύρια. Δεν πρέπει τα ζώα αυτά να βασανίζονται και να υποφέρουν οδεύοντας προς το θάνατο ούτως ή άλλως. Δεν είναι σωστό αυτό. Αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος. Πρέπει να συζητήσουμε για την ε, υπόθεση αυτή το πώς βλάπτεται και εξαπατείται και ο καταναλωτής με τις υποθέσεις αυτές, γιατί είναι σαφές πως ε, το άγχος ε, της μεταφοράς ε, δεν είναι καλό και για το κρέας τελικά που παράγεται από αυτή τη διαδικασία. Τι νόημα έχει δηλαδή. Το είπατε κι εσείς μόνο σας κύριε εισηγητά, να ξεκινάνε από την Ολλανδία και τη Δανία και να πηγα... τα χοιρινά και να πηγαίνουν στην, στην Πάρμα και να φτιάχνουμε μετά το περίφημο το προσούτο. Άμα, ήθελα, άμα θέλω προσούτο, θέλω ε, να είναι ντόπιο πραγματικά 100%. Είναι δηλαδή εξαπάτηση των καταναλωτών. Ε, αυτά τελικά δεν εξυπηρετούν την ε, ευρωπαϊκή οικονομία, βλάπτεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην, ε, στα προϊόντα αυτά. Υπάρχουν λοιπόν για μένα πάρα πολλοί λόγοι για τον κανονισμό αυτών ε, των 8 ώρων. Είπατε 37% μεταφέρονται σε περισσότερες από 8 ώρες. Σας πιστεύω. Αλλά θεωρώ πως ε, τότε είναι 37% παραπάνω ε, από όσα πρέπει. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, μια που λείπει η γητριά μας, θα ήθελα εγώ να παρουσιάσω σύντομα την θέση της ομάδας μας. Πρώτα απ' όλα κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Βεβαίως για την άλλη οι κανόνες μεταφοράς των ζώων είναι πάρα πολύ σημαντικοί για να αγγιηθούμε μια σωστή μεταχείριση των ζώων ακόμα και όταν πάνε προσφαγή. Τώρα, διαβάζοντας την έκθεση είναι σαφές ε, πως ε, έχουμε κανόνες, ε, έχουμε τους αναγκαίους κανόνες, πρέπει απλά να εφαρμοστούν. Πρώτη παρατήρηση λοιπόν, τα μέτρα ελέγχου πρέπει να είναι καλύτερα. Αν είναι να έχουμε κοινού κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται κιόλα. Όταν πάνε τα ζώα προσφαγή ε, δεν μπορεί να θεωρούμε πως ε, μπορούμε και να τα μεταχειριζόμαστε όπως να είναι ή δεν μπορούμε να ακολουθούμε τους κανόνες και δεν πρέπει να ανεχθούμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο στην Ευρώπη όπου παράγουμε ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μεταφέρουμε σε τρίτες χώρες για σφαγή. Εκεί όπου δηλαδή δεν υπάρχουν ε, τόσο αυστηροί κανόνες προστασίας των ζώων. Τώρα, όταν μιλάμε για τη θέση της Άλτε για το 8ωρο αυτό. Έχουμε συναδέλφους που λένε πως ε, πρέπει να επιμείνουμε σε αυτόν τον κανόνα, άλλοι λένε πως θα πρέπει ίσως ε, να τεθεί ένα μάξιμουμ ή ένα minimum. Ίσως να χρησιμοποιηθεί κάποια νέα τεχνολογία γι' αυτό. Άλλοι λένε πως ε, ο κανόνας αυτός ε, του οχτάωρου δεν είναι λογικός ε, και πρακτικός ε, δεδομένου παραδείγματος χάρη του ότι κάποια ζώα πρέπει να μεταφερθούν δια θαλάσσης. Και δεν είναι πρακτικός άρα αυτός ο κανόνας. Και κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν πως συνθήκες μεταφοράς είναι σημαντικότερε από το 8ωρο, το εάν ταΐζονται παραδείγματο χάρη τα ζώα. Οπότε η ομάδα μα δεν έχει κάποια ξεκάθαρη θέση. Κάποιοι συνάδελφοι ψηφίζουν έτσι, κάποιοι συνάδελφοι αλλιώ στην ομάδα μας. Οπότε θα πρέπει να αποφασίσουμε στη ψηφοφορία. Δεν έχουμε εδώ πέρα εμεί ξεκάθαρε ε, κόκκινε γραμμέ επί της αρχής στηρίζουμε τους ξεκάθαρους κανόνες που θα επιβάλλονται όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με λίγο νεράκι γιατί και εγώ έχω διψάσει σαν ε, άλογο. Εντάξει. Um, um, Είμαι σκιώδης εισηγητής, λοιπόν, σε αυτό το θέμα και σε ένα μεγάλο βαθμό συμφωνώ με τα όσα συμπεριλαμβάνει η έκθεση. Εδώ είχαμε να κάνουμε όχι τόσο πολύ με την ευζοία των ζώων, αλλά με την μεταφορά αυτών. Και αυτό δεν ήταν απλώς ε, η αιτιολόγηση, ήταν ένα γεγονός. Όμως, προς τον εισηγητή, πρέπει να πω ότι η ομάδα μου, η πράσινη, θέλουν με κάθε τρόπο να βρεθεί συμφωνία. Εδώ λοιπόν, μας είπε ο εισηγητής ότι ενώ συμφώνησε με πολλέ από τι τροπολογίε, τελείω συντοματικά φαίνεται να μην συμφώνησε με καμία από αυτέ των πρασίνων. Το οποίο εμένα με λυπεί. Συνάδελφοι, δεν μιλάμε για την ε, μεταφορά τούβλων ή ασβεστόλιθου. Μιλάμε για όντα που αισθάνονται, αναπνέουν, ε, συναισθάνονται και μπορούν να αισθανθούν τον πόνο και το άγχος. Είναι πολύ απλουστευτικό να πιστεύουμε ότι Ε, μπορούμε εμείς ως πλέον προηγμένο είδος να λύσουμε το θέμα αυτό με τρόπο υπεύθυνο. Και αυτό, επειδή προσωπώ την νοτιοανατολική Αγγλία και το μόνο λιμένα της χώρας όπου επιτρέπεται η εξαγωγή ζών των ζώων προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα, αυτό λοιπόν είναι πολύ ευαίσθητο για μένα. Και είναι και κάτι που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ έχω πάει στο λιμένα αυτό, έχω γνωρίσει τους κτηνοτρόφους, τους ε, ανθρώπους που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ε, ζώων. Έχω συναντήσει προσώπους με κυβερνητικών οργανώσεων, κτηνοτρόφους, εξαγωγής προϊόντων. Ξέρω ακριβώς ποια θέση θέλω να περάσει εδώ. Ξέρω γιατί έχω την άποψη που έχω, γι' αυτό και υποστήριξα την γραπτή δήλωση για τα συγκεκριμένα όρια και αυτό είναι ζήτημα απογορευτικό, κόκκινο, κόκκινη γραμμή για τους πρασίνους δεν φαίνεται ότι μπορούμε να επιτύχουμε κάποια συμφωνία, όμως εμείς με κάθε τρόπο θα θέλαμε να επιτευχθεί αυτή. Να βρούμε βεβαίως συνεννόησεις, να συνεργαστούμε και ελπίζω πραγματικά ότι ο εισηγητής θα μπορούσε να εξεύρει συμβαστικές τροπολογίες που θα λάβουν υπόψη το γεγονός ότι δεν μιλούμε για άψυχα δικείμενα. Ομιλούμε για ζώα. Ομιλούμε για την ανάγκη να μεταφέρονται σε όσο το δυνατόν μικρότερες αποστάσεις. Με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους. Ταξιδεύουν για να μετατραπούν σε τρόφιμα. Ε, τουλάχιστον να πηγαίνουν κοντά στο μέρος που μεγάλωσαν. Ελπίζω λοιπόν ο εισηγητής να έχει κάποιες ε, πρωτότυπες, νέες ιδέες, ώστε να καλύπτονται και αυτές τις προτεραιότητες. Σας εξηγώ ότι τις ε, ευαισθητοποιούν πολλοί κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Η κυρία Φώστερ, για τους αστυνομικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, με συγχωρείτε συναδελφοί, έχασα την αρχή της συζήτησης, διότι άλλαξε κάπως το ωράριο για σήμερα το απόγευμα. Δεν θα μιλήσω εκ μέρους του κ. Βαντόλεν, ε, που είναι ο σκιώδης εισηγητής γιατί από την δική μα την ομάδα θα συμφωνούσαμε με τι τροπολογίε, τι περισσότερε τροπολογίε Όμως θέλω να μιλήσω ω αντιπρόεδρος της ε, διακομματική ομάδα για την ε, ευζοία των ζώων και ω Βρετανή συνάδελφο. Τη συζήτηση αυτή την κάνουμε εδώ και 10 χρόνια. Το βρίσκω τραγικό αυτό. Και όπω είπατε και εσεί πρόεδρε και κάποιοι συνάδελφοι που είναι μέλη τη Επιτροπής αυτή επί χρόνια, τα έχουμε ξανασυζητήσει την υποχρέωση των οδηγών, ε, όλε αυτέ τι λεπτομέρειε, όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να βρούμε κάποιες λύσεις και όπως ο συνάδελφος ε, των Πρασίνων και εγώ συμφώνησα με την οκτάωρη μεταφορά. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Στα Σετλάντζ, ας πούμε μπορεί να μην είναι απλό να περάσει ένα ζώο από νησί προς την ενδοχώρα. Όλα αυτά πρέπει να λεφθούν υπόψη. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν και κάποιε αιτιολογημένε, μετρήσιμε εξαιρέσει. Νομίζω πάντω το συμπέρασμα είναι και για του σκοπού τη Επιτροπή αυτή, όπω σωστά και εσεί το θέσατε, είναι ότι το θέμα ανάγεται σε μείζον λόγω των κανόνων που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από κάποια χρόνια για τα σφαγεία. Γι' αυτό ακριβώ κάποια ζώα μεταφέρονται για μεγαλύτερε αποστάσει ε, ανά την Ευρώπη. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι θα υπάρξει σοβαρή βελτίωση αν δεν υπάρξει και σοβαρή αλλαγή της φιλοσοφίας μας για το πού πρέπει να θανατώνονται τα ζώα. Εάν θέλουμε καλή ζωοτεχνική μέθοδο, εάν θέλουμε να υπάρξει πρόοδος και εδώ, είναι ένα από τα μείζωνα ζητήματα που θα πρέπει να λύσουμε. Μην ξεχνάμε και τη μεταφορά των ζώων που πηγαίνουν από την Ανατολική Ευρώπη πολλές φορές για να καταλήξουν στη Σικελία πόσο κοντά είναι αυτό στην πηγή. Εδώ λοιπόν κάποιε από τι τροπολογίες σίγουρα είναι θετικέ, θα τι στηρίξουμε, αλλά είναι και άλλες οι αρμόδιες επιτροπές και αυτό που θέλουμε είναι να πετύχουμε ένα χειρό μήνυμα. Έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε τα ζώα κατά τη μεταφορά τους και Βεβαίω είναι και ζώντα όντα τα οποία είναι μάλλον ζωντανά πλάσματα τα οποία έχουν τι απεριστήσει, αλλά μιλάμε και για εμπόρια εδώ και πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη. Ο κύριος Μπάχ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Λουίς Δεγκράντες Πασκουάλ για την έκθεσή του που έχει πάρα πολλά καλά σημεία, ειδικά την εναρμόνιση των μηχανισμών ελέγχου και την εκπαίδευση των οδηγών. Εδώ πέρα μπορούν να βελτιωθούν πάρα πολλά πράγματα. Και πως τα κράτη-μέλη πρέπει να ελεγχθούν ε, όσον αφορά τις, ε, τους ελέγχους και τις κυρώσεις που επιβάλλουν. Θεωρώ πως ο συνάδελφος Ντεγκράντες ε, εστιάστηκε στις ε, μεταφορές χωρίς να μπει σε συναισθηματικές πτυχές αλλά λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των ζώων. Και βεβαίως εδώ πέρα μπορούμε να είμαστε αρκετά θαραλέοι. Ο τίτλος ούτως ή άλλως το περιγράφει. Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Οπότε πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η πτυχή. Δεν είναι μόνο οι καταναλωτές που παρακολουθούν την υπόθεση αυτή, αλλά και όλοι οι δικοί μας λένε πως τα ζώα πρέπει να εκτρέφονται και να σφάγονται σε μικρές αποστάσεις. Δεν βλέπω και εγώ την ανάγκη γιατί να διασχίζουν ε, την Ευρώπη και να είναι 24 ώρες στον δρόμο για να σφαχτούν. Παρ' όλα αυτά, ευνόμαστε φιλόδοξοι και όπως είπαμε πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, μια αναλογικότητα μεταξύ οικονομικού συμφέροντος και προστασίας των ζώων. Νομίζω πως θα γίνει αυτό στη συζήτηση με τους κοιόδησίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Πριν από 15 χρόνια θυμάμαι πως έκανα καμπάνια υπέρ του να ισχύσουν οι τωρινοί κανόνες. Χρειάστηκαν κάποια χρόνια, αλλά τότε πολλοί άνθρωποι παράλογα ε, ζητούσαν ε, απαγόρευση εξαγωγών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τι θέλω να πω. Πρέπει να δούμε τα πράγματα λογικά και πρακτικά. Γιατί εάν τότε ακολουθούσαμε την κοινή γνώμη θα ήταν νόμιμο να διασχίσει κανείς ε, ολόκληρη τη χώρα, 15 ώρες ε, οδικός, αλλά θα ήταν παράνομο να περάσει ε, ένα ζώο το σύνορο στην, Ιρλανδία, στο ίδιο, σε ένα νησί πάνω μπορεί στην ίδια κατεύθυνση να οδηγηθούμε εδώ πέρα αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Οπότε έχω βάλει εδώ πέρα τι περιφερειακέ νήσου. Για να πάει κανεί ε, με καράβι στο Αμπερντίν από τι απομακρυσμένε νήσου χρειάζονται 12 ώρε. Οπότε σημασία έχουν οι συνθήκε, όχι πόση ώρα κάνει το καράβι. Γιατί υπό συνθήκες ε, ανάπαυσης ε, στο πλοίο και αυτό το οποίο συμβαίνει στο πλοίο είναι κατ' ουσίαν ε, μια περιοχή ανάπαυσης, ε, τότε δεν πρέπει να μετράει αυτός ο χρόνος. Αν επιμείνουμε οπωσδήποτε στι 8 οι ώρες, θα έχουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το, τα, οι Όρκνεϊ και Σέτλαντ δηλαδή θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αυτό το οποίο θα έλεγα επίσης για την ε, νομοθεσία για τα ασφαγεία. Επίσης, Έχουμε κάποιες τροπολογίες που εξετάζουμε. Ζητάνε να φύγει η διατύπωση για σφαγή. Εάν είναι δηλαδή να επιμείνουμε για το ίδιο όριο για ζώα που πάνε απλά από βοσκότοπο σε βοσκότοπο στη Βόρεια Ευρώπη. Κοιτάξτε, η διαχείμανση που λέμε ε, των κοπαδιών γίνεται εδώ και χιλιάδες χρόνια γιατί μπορούν να, να βόσκουν ε, τα ζώα το χειμώνα στη, Βόρεια Σκοτία και κατεβαίνουν στην Αγγλία. Και στη Σκανδιναβία το ίδιο. Δεν μπορεί να μεγαλώσει στο ίδιο μέρος ε, το ζώο και χρειάζονται και δυόμιση χρόνια ούτως ή για να γίνει ενήλικο το, το μοσχάρι. Οπότε εδώ πέρα απαγορεύεται η διαχείμανση. Τι κάνουμε τα, τα το βόρειο μέρος της Ευρώπης ε, τι θα βγει εκτός γεωργίας πρέπει να είμαστε λογικοί και να δούμε το τι βελτιώνει την ποιότητα ε, της μεταφοράς αντί να θέσουμε ένα απόλυτο όριο. Γι' αυτό υποστήριξα το 8ωρο ημερησίως με μια περίοδο ανάπαυσης πριν από τόσα χρόνια. Επίσης υπάρχει το ζήτημα της εκτροφής των ζώων. Πάλι, εάν αν φύγει η λέξη για σφαγή, τα ζώα υψηλή ποιότητας που πάνε για αναπαραγωγή κινούνται παγκοσμίω και θα βγει τελείω εκτός η Ευρώπη. Και το αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα θα είναι βεβαίως ε, μείωση τη ποιότητας ε, των, ε, των ζώων. Υπάρχουν πολύ καλέ προτάσει τώρα όσον αφορά τη βελτίωση των συνθήκων π.χ. εκπαίδευση των οδηγών, μέτρηση της ε, θερμοκρασίας ε, και τα λοιπά ε, εντός του φορτηγού, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες που δεν είναι καθόλου πρακτικές προτάσεις. δεν νομίζω πως μπορούν να μας βρουν σύμφωνος. Λίχτενμπεργκερ. Ναι, ζήτησα το λόγο. Γιατί για μένα δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ βελτίωσης της μεταφοράς περσέ και περιορισμού του χρόνου. Και τα δύο χρειάζονται εάν ε, παίρνουμε στα σοβαρά την προστασία των ζώων. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Όταν μιλάμε για τις συνθήκες μεταφοράς, ε, χρειάζεται μια επιτήρηση και χρειάζονται και υποδομές. Θα αναφέρω την υποδομή, γιατί εμείς στις Άλπεις διαπιστώνουμε ε, στο Μπρένερ, στο πέρασμα του Μπρένερ. Ε, υπήρξε, υπήρχε ένα σταθμός ε, μεταφόρτωσης ζώων που ταΐζονταν τα ζώα, ξεκουράζονταν. Και τι έγινε, το απέφευγαν οι ταλικέριδες για να μην υφίστανται ελέγχους. Γιατί βεβαίως έπρεπε και να πληρώσουν εκεί πέρα. Οπότε, όταν σταματούσαν κάποιον και διαπίστωναν υπέρβαση του χρόνου, έπρεπε να πάει τα ζώα εκεί πέρα και να αναπαυθούν τα ζώα, να ταϊστούν και τα Αυτή ήταν μια αποτελεσματική μέθοδος. Αυτά για, το, για αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό ε, δεν είναι κατά του χρόνου μεταφοράς γενικώ. Και άλλη μια εμπειρία μου. Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες γιατί λέτε ε, πως έχουν γίνει λιγότερα τα σφαγεία στις περιφέρειες. Μα υπάρχουν και κινητά σφαγεία σε κάποιες περιφέρειες, κάτι κοντέινερ εκεί πέρα, που περιέχουν μέσα ένα σφαγείο, που φροντίζουν ε, και τις μικρές απομονωμένες περιοχές. Γιατί δεν μπορούμε να ενισχύσουμε ε, αυτούς παραδείγματος χάρη για να αποφευχθεί τελείως η μεταφορά. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον αλλά αυτά δεν είναι επιχείρημα κατά του χρονικού περιορισμού, γιατί υπάρχουν αναγκαιότητες. Και έχουμε μια ευκαιρία να βελτιώσουμε την υγεία των ζώων. Γίνονται πολλές, πάρα πολλές μεταφορές και μια που μιλάμε για ζωντανά, πρέπει να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν πρόκειται για κοινέ μεταφορές. Ευχαριστώ να πω κι εγώ κάτι. Καταλαβαίνω αυτό το οποίο ακούστηκε για τους κανονισμούς όσον αφορά τα σφαγεία που επίσης φαίνεται πως αποτελεί πρόβλημα εδώ πέρα και σχετίζεται με τη μεταφορά ζώων ζώων γιατί εγώ θεωρώ πως τα ζώα πρέπει να σφάζονται όσο δυνατόν πιο κοντά στον τόπο αν αυτό σημαίνει σφαγείο στα Σέτλαντ, καλώς. Αλλά εξακολουθώ να θεωρώ πως οι αγρότες θα θένε να τα στέλνουν ζωντανά οπουδήποτε. Και όταν μπαίνει κανείς σε αυτή την κρίζα ζώνη, εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα. Γνωρίζω εγώ από τη δική μου την περιοχή πως κάποιες φορές ε, ο κανονισμός που ισχύει για τα σφαγεία προκαλεί περισσότερο Περισσότερο οδύνη στα ζώα από ό,τι πριν. Να δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα. Εάν ένα ζώο φτάσει τραυματισμένο στο σφαγείο, όχι άρρωστο, δεν μπορεί να σφαχθεί μέχρι να έρθει ο κτηνίατρος να πει πως είναι σε αρκετά καλή κατάσταση για να σφαγεί. Και αρχίζουμε να ψάχνουμε τον κτηνίατρο. Εν τω μεταξύ το ζώο υποφέρει. Πονάει το ζώο, αλλά ο κανονισμός λέει πως πρέπει να το βγάλει ο κτηνίατρος υγιές για να σφαγεί. Καταλαβαίνω όταν είναι άρρωστο το ζώο να μην περάσει στην τροφική αλυσίδα, αλλά άμα του έχει σπάσει το πόδι, μου φαίνεται χαζό το σύστημα εδώ πέρα. Εγώ είμαι υπέρ του 8 Γιατί είμαι απογοητευμένος. Γιατί. Λόγω των 20 τόσων ετών που είμαι σε αυτό το κοινοβούλιο προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για την μεταφορά ζών των ζώων. Και αποτύχαμε. Η αποτυχία μπορεί να οφείλεται όχι οπωσδήποτε στους κανονισμούς, αλλά μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν ε, εφαρμόζονται. Και υπάρχει υπάρχει μία έτσι νοοτροπία, ας γίνει ό,τι γίνει. Ε, και πώς συμπεριφέρονται οι μεταφορές στα ζώα. Αλλά, όπως είπε ο κύριος ε, Τέιλορ, είναι μεγάλο το ζήτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα περισσότερα email που λαμβάνουμε αφορούν τα ζώα. Τώρα το αν αντικατοπτρίζει αυτό την αγγλική κοινωνία δεν θέλω να το σχολιάσω, αλλά είναι γεγονός. Είναι γεγονός. και εξάπτονται έτσι τα συναισθήματα των Βρετανών ε, βουλευτών. Συμφωνώ λοιπόν με το αίτημα του κυρίου Ντεγκράντες για να αναβληθεί η ψηφοφορία για να προσπαθήσουμε να, να συμφωνήσουμε. Αλλά συμφωνώ μαζί του επίσης πως εάν μέχρι τις 7 Μαΐου δεν γίνει τίποτα θα τεθεί σε ψηφοφορία και τι γίνει. Η ειρωνία είναι εγώ είμαι αναπληρωτής δε στην Επιτροπή Γεωργίας και όταν το μάθουν εκεί πέρα, ο Θεός να μας βοηθήσει. Γιατί αν έχει κάποιο συμφέρον είναι αυτή η Επιτροπή. Αλλά ε, τι να κάνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Α δούμε τώρα. Εγώ θα ζητήσω από τον εισηγητή και τους κοιόδους εισηγητές να προσπαθήσουν να συνεργαστούν, να βρουν ε, συμβαστικές τροπολογίες. Εάν όχι θα αναβάλουμε τη ψηφοφορία και ό,τι γίνει. Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών. Ποιος είναι. Νόργκρουμ ή Ανιέλη. Well, I assume that must be Mr. Giavinelli. Yeah. Υποθέτω ότι είστε ο κύριος Τζαβινέλη. Ε? Ποιος... Ε, για κυρία δεν μου φαίνεστε δηλαδή, πώς να το πω. Έχετε το λόγο, εν πάση Ε, <clears throat> ε, Καλησπέρα σα είμαι ο Αντρέα Γκαβινέλη, υπεύθυνο της γενική διεύθυνση ΣΑΝΚΟ για την ευζοία των ζώων. Ευχαριστώ την Επιτροπή σα που ασχολείται με το θέμα τη μεταφορά των ζώων και, για τα σχόλια που μα αποστήλατε. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναλαμβάνω ότι παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τι εργασίε του Κοινοβουλίου και βεβαίω τι σχετικέ συζητήσει και στο Συμβούλιο. Και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σημαντικό να εργαστούμε ώστε να βελτιώσουμε την εφαρμογή του κανονισμού περί των μεταφορών όπου βάσει των διαθέσιμων σημερινών στοιχείων η μεταφορά των ζώων στην Ευρώπη είναι μια πραγματικότητα και από το 2005 ως σήμερα, όπως επιβεβαιώνει και η σχετική έκθεση της Επιτροπής, υπήρξε και αύξηση της μεταφοράς ζώων. Άρα πρόκειται για μια προτεραιότητα. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι μεταφέρονται τα ζώα σε συνθήκες καλής, ε, μάλλον ευζωίας και καλής υγείας. Όπως το ζητούν και οι πολίτες. Βεβαίω, σε σχέση με όσο αναφέρθηκαν εδώ, το όλο ζήτημα για τις, των οκτώ η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά είναι η ίδια με αυτή που αναφέρεται και στην έκθεση που δημοσιεύτηκε. Σε αυτή τη φάση δεν επιδιώκουμε τροποποίηση του κανονισμού, αναθεώρηση δηλαδή των κανόνων σε σχέση με το χρόνο μεταφοράς, τη διάρκεια μεταφοράς, αλλά δεσμευόμαστε να αποτιμήσουμε σχετικές προτάσεις ώστε το σύστημα της ε, δορυφορικής πλοήγησης, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, να χρησιμοποιηθεί κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, όπως και το σύστημα συλλογής πληροφοριών για τους ελέγχους που διεξάγουν τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η δύο βραχυπρόθεσμοι στόχοι μας, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη και εδώ να σας ενημερώσω ότι έχουμε και την πρόθεση να αποτιμήσουμε και τις προτάσεις του Κοινοβουλίου, ποιες και αν είναι αυτές, και οπωσδήποτε να επιδιώξουμε και τον περιορισμό του διοικητικού άχθους ώστε να υπάρξει και καλύτερη χρήση των ε, τεχνολογιών ηλεκτρονικής συχνηλεξιμότητας. Αυτή είναι η στόχη που έχουμε θέσει και ευχαριστώ και πάλι την Επιτροπή σας για το έργο της. Ευχαριστώ. Κύριε Ντεγκράντες, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ, κύριε Σίμψον. Σύντομο. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω τις θέσεις. Πρώτον, όλοι, επιμένω, είμαστε υπέρ της καλής μεταχείρισης των ζώων. Όλοι. Είναι προφανές αυτό. Και εννοείται μας τιμά όλους. Δεύτερον, ποια είναι η πραγματικότητα. Πώς θα βελτιώσουμε την καλή μεταχείριση των ζώων κατά την μεταφορά τους. Αυτό μας απασχολεί στη γνωμοδότηση αυτή που έχουμε μπροστά μας. Δεν θα ήταν φυσιολογικό η Επιτροπή Μεταφορών που γνωμοδοτεί να κάνει κάτι διαφορετικό από το να αναφερθεί στις μεταφορές. Κύριε Τέιλορ, αυτό που μας απασχολεί είναι το ζώο, η μεταφορά του, αλλά εφόσον είμαστε Επιτροπή Μεταφορών πρέπει να εξετάσουμε την οπτική γωνία της μεταφοράς. Τι λύσεις μπορούμε να βρούμε για την μεταφορά. Επιμένω λοιπόν ότι από τις συζητήσεις που έκανα με τους Σκιώδης δεν υπάρχουν άλυτα προβλήματα. Εκτός από ένα που είναι εκείνο των οκτώ ωρών. Δεν βλέπω να συμφωνούμε πάνω σε αυτό. Κατά τα άλλα, ναι, πιστεύω ότι είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε. Με κατηγορείτε κατά κάποιο τρόπο ότι δεν έχω λάβει υπόψη μου καμία από τις τροπολογίες σας. Ναι, αλλά από τις τροπολογίες σας θα φτιάξω μεταξύ άλλων τις συμβαστικές μου. Δηλαδή θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω το πνεύμα το οποίο περιλαμβάνεται στις τροπολογίες σας. Και ευχαρίστω να υποβάλλετε και άλλες. Το θέμα είναι να μην συμπεριφερόμαστε ριζοσπαστικά και να βρούμε μία λύση που να μας ικανοποιεί όλους δεν γίνεται. Υπάρχουν συμφέροντα απόλυτα θεμητά και υπάρχουν και διαφορετικές συνθήκες. Μιλήσατε για τα νησιά. Ε, πράγματι, δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, αλλιώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της θαλάσσιας μεταφοράς από ότι της οδικής. Οι αποστάσεις είναι αυτές που είναι, δεν μπορούμε να τις κόψουμε, να τις μικρύνουμε. Τα νησιά βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Ε, και με εμά το ίδιο είναι. εμεί επίση έχουμε τα νησιά με τι χελώνες μα. Συνεπώς, δεν υπάρχει τέλεια λύση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξαιρέσεις και ειδικέ περιπτώσεις. Ως Επιτροπή Μεταφορών όμως, έτσι κι Δεν μα ζητούν τόσο πολλά πράγματα. Επί τη ουσία αρμόδια είναι η Επιτροπή Γεωργίας. Εκείνη προσπαθεί να βρει ελαστικές λύσεις. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι το 8 αποτελεί σημείο αναφορά. Είναι ένα σημείο αναφορά αλλά δεν θα πρέπει να είναι κάτι το άκαμπτο, το οποίο να μην επιδέχεται στις μεταφορές ε, τίποτα άλλο. Γιατί όπως είπαμε υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα επειδή είναι διαφορετικές οι περιφέρειες στην Ευρώπη. Κύριε Σίμψον, θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία μέχρι τις 7 Μαΐου. Για το 8ωρο, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα βρεθεί κανένας τρόπος να συμφωνήσουμε όλοι. Όμως, αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε επί της ουσίας και δεσμεύομαι, Πρόεδρε, να συνεχίσω να δουλεύω με τους κοιόδης εισηγητές και με τους ε, εισηγητές και με σας ε, τον ίδιο κύριε Πρόεδρε που εννοείται ότι και εσείς πρέπει να μας πείτε την γνώμη σας και θα την σημειώσουμε. Και ελπίζω ότι θα μπορέσω να παρουσιάσω κάτι που να μας βρίσκει όλους πολύ κοντά. Ακόμα και αν δεν συμφωνήσουμε με όλα. Τέλος, να ξέρετε ότι αντιλαμβάνομαι όλες τις αποχρώσεις που ακούσαμε και θα προσπαθήσω να πετύχω κάποια συμφωνία για την 7η Μαΐου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Τεγκράντες. Όντω αναβάλλεται για την 7η Μαΐου η ψηφοφορία. Οπότε, ελπίζω να καταφέρουμε μέχρι τότε να έχουμε πετύχει συμφωνία. Αλλιώς, απλώς θα ψηφίσουμε και θα δούμε τι θα βγει από την ψηφοφορία. Ο εισηγητή και οι σκιώδες θα πρέπει να βρεθούν να συζητήσουν και να προσπαθήσουν να πετύχουμε λύση επόμενο θέμα είναι η στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγγήτρια βγήκε. Σε δύο λεπτά θα είναι πίσω, μου λένε. Φοβερό.

Έφτασε η κυρία Τικάου, έκανε ένα sprint, δεν ξέρω από πού. Πολιτική συνοχή για την περιοχή του Ατλαντικού είναι το θέμα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη που άργησα αλλά βλέπετε ήμουνα στην Ήτρε, στην συνεδρίαση εκεί. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την Γραμματεία και όλους τους συναδέρφους που με βοήθησαν να ετοιμάσω τη γνωμοδότηση αυτή. Θέλω σύντομα να σας μεταφέρω κάποια πράγματα από την γνωμοδότηση αυτή. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει σχέδιο δράσης για την στρατηγική μας όσον αφορά τον Ατλαντικό μέχρι το 2013 εισαγάγοντας προγράμματα τα οποία να είναι τέτοια ώστε να αποφελούνται όλες οι πλευρές. Η γνωμοδότηση αυτή μιλάει για την μεγάλη σημασία που έχει η θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό και ενθαρρύνει τους ε, εταίρους να συμμετέχουν στο σχετικό φόρουμ όταν αυτό χρειάζεται. Θέλουμε επίσης ένα πολύπλευρο σύστημα στην περιοχή του Ατλαντικού. Είναι αναγκαίο κάτι τέτοιο. Και πρέπει να επικεντρωθούμε και στον βόρειο άξονα και στον ε, νοτιοδυτικό. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τους ε, μηχανισμούς διασύνδεσης. Πρέπει επίσης να δώσουμε μεγάλη σημασία στη σύνδεση μεταξύ των λιμένων και των εσωτερικών οδών των πλωτών ώστε ολόκληρη η περιοχή να μπορεί να αποφεληθεί από τις θαλάσσιες μεταφορές. Αναγνωρίζουμε ότι έχει μεγάλη σημασία ε, και έχουν μεγάλη σημασία και οι εμπορικές μεταφορές, όπως ε, επίσης ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέρη της περιφέρειας θα αποφεληθούν ε, μας ενδιαφέρουν επίσης οι μικρής απόστασης μεταφορές. Πιστεύουμε ότι έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα το περιβάλλον και ζητούμε από τις αρχές των χωρών να υπογράψουν ένα μνημόνιο κατανόησης για να ε, μειωθεί η συμφόρηση του δικτύου και να υπάρξει καλός έλεγχος των θαλάσσιων μεταφορών. Υπογράψουν επίσης συμφωνία για ανταλλαγές ε, δεδομένων όσον αφορά τις μεταφορές αυτές και να καταπολεμηθεί το διασυνοριακό έγκλημα. Θέλουμε επίσης να εφαρμοστούν και προγράμματα όπως είναι το έγνος και το γαλιλαίο, προκειμένου να καλυφθούν τα υποστηρικτά συστήματα έρευνας και διάσωσης του Ατλαντικού. Τονίζουμε επίσης την ανάγκη για παρετέρω ανάπτυξη του τουρισμού Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω πόσο μεγάλη σημασία έχει παρετέρω ανάπτυξη στο μέλλον των κύριων στοιχείων της Ατλαντικής περιοχής, όπως είναι οι θαλάσσιες μεταφορές, ναυσιπλοεία, η δατοκαλλιέργεια, η αλία, ο τουρισμός, η ενέργεια από τη θάλασσα και άλλοι δρόμοι για την προμήθεια ενέργειας. Πρέπει όμως να σας πω ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωσή της δεν είναι τόσο συγκεκριμένη όσο εμείς θα επιθυμούσαμε για μια τέτοια στρατηγική. Και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν διαθέτει σχέδιο δράσης. Ζητάμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλη του 2013 να μας έχουν παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης το οποίο να περιλαμβάνει όλους τους φορείς της περιοχής, όλους τους εταίρους στην περιοχή και να φροντίσει να βελτιωθεί η κατάσταση στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ πολύ όσον αφορά τι μεταφορές. Ευχαριστώ. Σε για το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να συγχαρώ την συνάδελφο για την εξαιρετική τη δουλειά. Όπως συνήθως βέβαια, όποτε αναλαμβάνει κάποιο θέμα, τα πλαίσια της Επιτροπής μας σε καιρούς ε, πίεσης ε, δημοσιονομικής, λιτότητας και χρηματοπιστωτικής κρίσης αναζητούμε λύσεις που να επιτρέψουν την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μια δεσμή μέτρων για να τονώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και θα πρέπει ακριβώ και τα κράτη-μέλη να οργανώσουν έτσι τι πολιτικέ του ώστε να εκμεταλλευτούν τι ευκαιρίε που παρουσιάζει η πράσινη οικονομία. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι θα πρέπει να στραφούμε και προ τη θάλασσα. Να την εξετάσουμε την περιοχή, την ε, περίπτωση αυτή και να σκεφτούμε και τη γαλάζια οικονομία που μπορεί να μας επιτρέψει να επιδιώξουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας. Ήθελα λοιπόν κάποια σύντομα σχόλια να κάνω ως προς τα βασικά σημεία της ε, έκθεσης. Πρώτα απ' όλα, συγχαίρω για τη συμπερίληψη της μνήας των θαλάσσιων αυτοκινητοδρόμων και των λιμένων, αλλά με κάποια δυσαρέσκεια βλέπω ότι η μνήα αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στους ανάλογους προσανατολισμούς των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς, ούτε στη διευκόλυνση σύνδετας στην Ευρώπη. Connecting Europe. Θα έπρεπε να ενισχύσουμε ακόμη την σημασία τη τόνωση των επαγγελματικών κλάδων που έχουν σχέση με την θάλασσα. Σε πολλού τομεί χρειάζονται επαγγελματικά προσόντα όπω την αυπηγία, τον ε, ε, θαλάσσιο τουρισμό και την αλεία στρατηγική για τον Ατλαντικό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιφερειακούς, τοπικούς και εθνικούς φορεί. και ήδη θα έπρεπε να έχει υποβληθεί μια σχετική πορεία από το 2010 και όχι από το 2014 όπως αναφέρεται. Επίσης λειτουργικά προγράμματα που σχετίζονται με τα διευθυντικά ταμεία και προέρχονται από τα διευθυντικά ταμεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να σχεδιαστούν πριν το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Τέλο, ε, αλλά δεν είναι λιγότερο σοβαρό αυτό το σχόλιο, η εξωτερική διάσταση της στατική αυτής για τις υπερπόντιες περιοχές είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουν και αυτές να στηριχθούν. Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 60% ε, της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης βασίζεται στα ε, στα υπερπόντια διαμερίσματα, 15.000 20.000 συνολικά τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, το πώς λειτουργούν αυτές οι οικονομίες που βασίζονται στη θάλασσα, εκμεταλλευόμενοι την ενέργεια, την ενέργεια που μπορεί να σχετίζεται με την, ε, να παράγεται μέσα από τη θάλασσα, τις ναυτικές δραστηριότητες, καθώ και την επιστημιστική ασφάλεια. Πρέπει να σκεφτούμε την πρόσβαση των περιοχών αυτών στην ενιαία αγορά και σε όλε τι δυνατότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιδιώξουμε κατά αυτόν τον τρόπο του στόχου μα. Θέλω να συνεργαστώ ε, και να δηλώσω εδώ την προθυμία μου ε, για επικοδομητική ακριβώ προσέγγιση και με την εισηγήτρια και με του κέντρου εισηγητέ, προκειμένου να εξεύρουμε μια ικανοποιητική λύση για την ε, στρατηγική αυτή. Κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Μπιλμπάο δεν ήρθε. Ήταν σημαντικό να μιλήσει, αλλά θα τα μιλήσω εγώ. Ευχαριστούμε την κυρία Τσικά για την ως συνήθως εξαιρετική δουλειά της. Κάτω το δεν βλέπω εγώ εδώ πέρα είναι οι αεροπορικές συγκοινωνίες. Νομίζω πως ε, κολλάνε εδώ πέρα και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά παραπέρα γιατί αν μιλάμε για τον Ατλαντικό εντάξει καλά είναι και τα λιμάνια και την ε, παράκτια ναυτιλία, αλλά το θέμα είναι αν έχετε δει, παραδείγματος χάρη, τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Το είπε, νομίζω, το είπε και ο συνάρφος ο οποίος προηγήθηκε. Αλλιώς συμφωνούμε με την ε, κοινή χρήση δεδομένων, καταπολέμηση των δυσκολιών, ε, πολλά από αυτά τα οποία περιέχονται στα άρθρα 7 και 8 και νέα με έκαναν να χαμογελάσω. Είναι θαλάσσια πολιτική. Ο Μπράιν Σίμψον θα μας πει πόσο σημαντική είναι αυτή η θαλάσσια πολιτική για να συνεχίσουμε σώμεθα και αυτό αφορά και πάρα πολλούς θαλάσσιους χώρους και τη Βαλτική και τη Μεσόγειο και το Ατλαντικό οπωσδήποτε. Υπάρχει μια μεγάλη γαλάζια ανάπτυξη η οποία θα επέλθει δηλαδή στην θαλάσσια η οικονομία και η Ευρώπη βεβαίως βρέχεται από τον Ατλαντικό και αυτό έχει σχέση και με τα θαλάσσια επαγγέλματα. Τα θαλάσσια επαγγέλματα δεν διαγράφτηκαν από εδώ μέσα γιατί λέτε πως δεν κολλάνε εδώ πέρα. Εγώ θεωρώ πως οπωσδήποτε ταιριάζουν σε αυτή την έκθεση και πρέπει να τα αναφέρουμε όταν μιλάμε και για στρατηγική ναυτιλία και όλα αυτά. Συνολικά λοιπόν μια καλή γνωμοδότηση δεν ξέρω τι θα συμπλήρωνε η κυρία Μπιλβάου. Οπωσδήποτε έχει κάποιες τροπολογίες, αλλά από όσο την ξέρω θα συμφωνούσα κι εγώ. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ο Τέιλορ για τους πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς θεωρούμε πως είναι εξαιρετική αυτή η έκθεση και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το ότι βλέπουμε κάποια στοιχεία διασυνοριακού συντονισμού, συνδέσει μεταξύ λιμένων και ενδοχώρας, ε, πλεύσιμα ποτάμια, των βασικών παραγόντων δε οικονομική ανάπτυξης και του ότι πρέπει να υπάρξει υψηλό ποιοτικό προϊόν, τουριστικό προϊόν, η ιδέα ενός σχεδίου δράσης για τον Ατλαντικό ε, είναι κάτι το εξαιρετικό και για να γίνει δε ο Ατλαντικός ε, μια περιοχή υπόδειγμα για την καθαρή ναυτιλία, όλα αυτά είναι στόχοι που εμείς επικροτούμε και θα καταθέσουμε και κάποιες ερωτάσεις. Α, να μένουμε βέβαια με επιτυχή κατάληξη. Η κυρία Φώστερ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Τσικάου, νομίζω πως κάλυψε πολλά θέματα θα συμφωνήσω με την κυρία Μάισνερ. Πρέπει να δούμε τον τομέα της αεροπορίας. Και αυτό κολλάει. Το ανέφερε, ανέφερε το έγνωση η κυρία Τσικάου και τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης. Αλλά νομίζω πως όλοι οι συνάδελφοι συνολικά έθεσαν ζητήματα με τα οποία συμφωνώ και ευχαριστούμε και την κυρία Τσικάου ως ομάδα. Κύριε Μπιλμπάου, συγγνώμη, προχωρήσαμε, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε. Αλλά τώρα ήρθατε και μπορείτε να μιλήσετε. Ευχαριστώ, έρχομαι από άλλη επιτροπή. Ήμουν και εκεί υπεύθυνη. Νόμιζα ότι θα πήγαινε αλλιώ το χρονοδιάγραμμα. Τέλο πάντων, ευχαριστώ πολύ την κυρία Τικαό για την έκθεσή τη. Πολύ σύντομα θέλω να σας πω ότι η έκθεσή της, η γνωμοδότησή της επικεντρώνεται πολύ στις λιμενικές δραστηριότητες και την βελτίωσή τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε εδώ και την ανάγκη να βελτιωθούν οι σιδηροδρομικές υποδομές, όπως επίσης και οι οδικές. Κάθε φορά να επιλέγεται η καλύτερη λύση για τη μεταφορά εμπορευμάτων πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνδέσεις που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να τα συνδέσουμε όλα αυτά και με άλλες εκθέσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν, το Europa Connecting και γενικότερα να το υπογραμμίσουμε αυτό, ότι δηλαδή πρέπει να συμπεριληφθούν και οι σιδηροδρομικές μεταφορές στην έκθεση αυτή για να επιμείνουμε στην ανάγκη που υπάρχει να αναπτύξουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα και σύστημα ποιότητας. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται μνήα στις διαφορετικές περιοχές ανάλογα με τους τρόπους μεταφοράς που χρησιμοποιούν. Επιμένετε πολύ στο θέμα των λιμένων, ενώ εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να αναφέρεστε και στα άλλα θέματα τα οποία σας είπα μόλις τώρα. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 38 ονόματα έχω εδώ. Δεν ξέρω. Εσείς. Ο κύριος Κίνγκ είναι... Α, ωραία. Εύκολο να το προφέρω. Πολύ πιο εύκολο από τα άλλα που βλέπω εδώ στον καταλογό μου. Παρακαλώ, εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν, ο κύριος Κίνγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επιτροπή που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε. Διαβάσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σχέδιο έκθεση. Περιέχει πολλέ αξιόλογε χρήσιμε προτάσει, τι οποίε θα εξετάσουμε. Θα εξετάσουμε προκειμένου να ετοιμάσουμε το πρόγραμμα δράσης μα. Η Επιτροπή ζήτησε να ετοιμαστεί ένα πρόγραμμα δράση όσο το δυνατόν συντομότερα. Στόχος είναι να είναι έτοιμο φέτος τον Νοέμβριο. Λαμβάνοντα υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις είναι δυνατόν. Ούτε μυστικό θα σα φανεί, ούτε θα εκπλαγείτε, λέγοντας ότι ο στόχος για τη στατική του Ατλαντικού ωκεανού είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη και οι περιφερειές τους θα μπορέσουν να σχεδιάσουν ε, με αρκετά τη μεγάλη χρονική απόσταση προγράμματα που να καλύπτονται από το δέσμη μέτρο του ορίζοντα 2020, τα διευθυντικά ταμεία, τα ταμεία συνεχή και το καθεξή. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη και τι περιφέρειε λοιπόν να θέσουν τι βασικέ επενδυτικέ του προτεραιότητε και τι ερευνητικέ του προτεραιότητε ε, πρόθεσμα και μετά να μπορούν να, να διαβουλευτούν κατά την περίοδο του καλοκαιριού δημοσίω να ακούσουμε λοιπόν και να αφουγκραστούμε τις ιδέες των καθομελών και των περιφερειών τους και κατά την υπόλοιπη χρονιά να οργανώσουμε στα ενδιαφερόμενα κατημέλη εκδηλώσεις και μαζί μέχρι τον Νοέμβριο να έχουμε ετοιμάσει πλέον ένα σχέδιο προγράμματος δράσης ώστε να ε, το εξετάσουμε και να εγκριθεί στο τέλος της χρονιάς. Για κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις να πω ότι από όσα υπόθηκαν και εμείς πιστεύουμε ότι το στοιχείο μεταφορών της του Ατλαντικού είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνον για την, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των λιμένων. Βεβαίως μπορεί να έχουν τεράστιο αντίκτυπο οι στην απασχόληση, στα ποσοστά της και στο να ενισχύσουν ε, από την άποψη των πόρων της παράκτησης οικονομίας. Μπορεί από εγκαταστάσεις offshore να φτάνει μέχρι και ενέργεια στις ακτές. Μπορεί να υπάρχει μεταφόρτωση εμπορευμάτων και εμπορική κίνηση. Προσπαθούμε όλα αυτά να τα αντικατοπτρίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, ενθαρρύνοντα τα κάτι μέλη να τηρήσουν θετική στάση Τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα που θα ζητήσουν να χρηματοδοτηθούν από το πακέτο χρηματοδότηση ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο, πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά την εθνικοποίηση τη Βεβαίως πρέπει να δούμε συνολικά τον Ατλαντικό ωκεανό, βεβαίως την ε, περιοχή μεταξύ Ανατολής και Δύσης και τις ε, υπερπόδειε περιοχές, αλλά και σε σχέση με τις ΗΠΑ και να λάβει και μια διεθνή διάσταση όλη αυτή η στρατηγική. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα προγράμματα που μπορεί να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2014 και κυρίως να δεσμεύσουμε και άλλους εταίρους, άλλες περιοχές εκτός Ένωσης για την προώθηση αυτής της στρατηγικής. Σκοπός εδώ βεβαίως είναι η ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας στις θαλάσσιες, τις ε, παράκτιες οικονομίες, ε, γαλάζιες οικονομίε, γαλάζιε θέσει εργασία, όχι μόνο με τη χρήση κρατικών κονδυλίων, αλλά και με την ε, ιδιωτική συμμετοχή δυνατών. Θέλουμε εύστοχα, εύστοχα και χρήσιμα προγράμματα ε, που θα κατασκευάσουν τα κρατημέλη να προτείνουν μάλλον τα κρατημέλη να εξυπηρετούν τι ανάγκε αυτών των ε, απομακρυσμένων περιοχών. Και έτσι, εφόσον τεθούν επιτάπητο, να προκύψει και η χρηματοδότηση από τώρα στο 2020. Αυτό είναι ο απότερο σκοπό μα. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ την Επιτροπή για τη συνεισφορά τη και πραγματικά βρίσκουμε ότι είναι και πολύ χρήσιμη και πολύ αξιολογή. Θα φροντίσουμε λοιπόν σε συνεργασία με τα κρατημέλη να ετοιμαστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα δράση που να απηχεί τι προτεραιότητε που και εσεί μα επισημάνατε. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ανυπομονούμε λοιπόν να σα δούμε στο Λίβερπουλ και στο λιμάνι του, κύριε πρόσωπε τη Επιτροπή. Κυρία Τικάου, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για τι παρεμβάσει του. Ανυπομονώ και εγώ να δω τι τροπολογίε σα και μπορείτε να υπολογίζετε στη δική μου την ε, συνεισφορά. Συμφωνώ ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις διατάξεις που αφορούν τις υδροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές. Δυστυχώς Υπήρξε κάποιος περιορισμός στον αριθμό των χαρακτήρων, έτσι, το γνωρίζετε όλοι αυτό. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τον αριθμό λέξεων που θα χρησιμοποιηθούν, οπότε δεν μπορούσαμε να τα καλύψουμε και όλα. Ολοκληρώνοντας πάντως να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για τη στήριξή της και βεβαίως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Πνεύμα Συνεργασίας που επιδεικνύει. Έχω μια ερώτηση. Δεν είμαι βέβαια εάν κατανόησα σωστά Εξ όσων λοιπόν κατάλαβα, πρόγραμμα δράση, μάλλον σχέδιο πρόγραμματο δράση, θα ετοιμαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να υποβληθεί σε δημόσιε διαβουλεύσει πριν το τέλο τη χρονιά. Σωστά. Το σχέδιο προγράμματος δράσης όμως ή το τελικό κείμενο θα είναι έτοιμο το τέλος της χρονιάς. Ε, αν λάβω υπόψη τι κλασικέ απαντήσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λένε Νοέμβριο, αλλά εννοούν στην καλύτερη περίπτωση στο τέλο τη χρονιά. Θέλετε όμω να απαντήσετε σε αυτό, κύριε Κίνγκ. Ναι, για να είμαστε απολύτω σαφεί. Πρόγραμμα δράση, σχέδιο πρόγραμματο δράση, Νοέμβριο 2012 θα έχουμε. Και το τελικό κείμενο. Ελπίζουμε ότι το φόρουμ του Ατλαντικού θα ολοκληρώσει τι διαβουλεύσει του τον το νωρίτερο το Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2013. Οπότε θα επιδιώξουμε έγκριση, τέλο πάντων, ε, την έγκριση του προγράμματο δράση μέχρι τον Μάρτιο του 2013. Ωραία. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 7 Μαου. 13 Μαΐου συζήτηση στην Επιτροπή. Επιτροπή Περιφερειών ψηφίζει 31 Ιουνίου σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και την κυρία Τσικάου και την κυρία Μπιλμπάου που έτρεξαν και ήρθαν εδώ γέρος. Τώρα θα περάσουμε στη συνάντηση των συντονιστών.